Είναι όλα τα πρόσωπα χαρούμενα. Φανταστικό. Δυστυχώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Πρέπει να συζητήσουμε σήμερα το πρωί για κάτι που αποφασίσαμε χτε. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Δεν θέλω να τα λέω αγγλικά. Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ σωστή. Εχθέ ε, είχαμε τη συνεδρία των συντονιστών και αποφασίσαμε, το πήρατε με email, η για τη συνεδρίαση στο Ναϊρόμπι, η δεύτερη, δική μας, να είναι η Σαμπίνε Φερχάιν. Η Μαρία Μπαντία επί σειρά ετών, τρία χρόνια νομίζω, μας εκπροσωπούσε και η Σαμπίνε Φερχάιν είναι μαζί της τώρα σε αυτό το πράγμα, πώς το λένε, ε, διακυβέρνηση από το διαδίκτυο. Ένα φόρουμ που γίνεται για τη διαδικτυακή διακυβέρνηση και όπως ξέρετε πάει αυτό στο Ναϊρόμπι. Αποφάσισε το Προεδρείο όμω ότι πρέπει να, μπορούν να πάνε μόνο δύο. Ε, δύο ήταν από την Ήτρε, από την Επιτροπή Βιομηχανία και μία εκπρόσωπο από εμά. Εχθές το βράδυ λοιπόν είδα τα έγγραφα που λένε ότι έχει δύο έδρες το ΕΛΚ και τη μία την πήρε μια βουλευτής του ΕΛΚ, Ισπανίδα. Η δεύτερη έδρα ήταν ελεύθερη. Και χτες το βράδυ θεωρούσαμε ότι επειδή οι σοσιαλιστέ, μάλλον οι σοσιαλιστές ε, τηρούσαν στάση αναμονή και περίμεναν να δουν τι θα κάνουμε εμεί. Γι' αυτό δεν κάλυψαν τη θέση. Και αποφασίσαμε όχι αποφασίσαμε, ψηφίσαμε δηλαδή, Εχθέ το βράδυ, ψηφίσαμε και ορίσαμε τη Σαμπίνε Φερχάιν ω δική μα εκπρόσωπο τη Επιτροπή Πολιτισμού για το Φόρουμ τη Ηλεκτρονικής διακυβέρνηση. Σήμερα το πρωί λαμβάνω μια επιστολή από τον κύριο Ρόιλ που δυστυχώς την έστειλε αργά και που κανονικά δεν θα έπρεπε να τη στείλει με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν υπήρχαν τα έγγραφα. Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου αποφάσισε που την έχω εδώ. Το Κοινοβούλιο, το Προεδρείο αποφάσισε τα εξής και τα διαβάζω κατ' εξαίρεση αποφασίσε και κατόπιν αιτήματο των πολιτικών ομάδων υπό το φω της πολιτικής σημασίας του γεγονότος να εγκρίνει μία αντιπροσωπεία ad hoc τρίμελη η οποία θα οριστεί μετά από συμφωνία των Επιτροπών Βιομηχανίας και Πολιτισμού και η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει και ένα μέλος της ΣΤΟΑ. Και έρχομαι τώρα ε, στον κύριο Ρόιλ, τον πρόεδρο τη Άλλη Επιτροπή, όχι possibly ενδεχομένω, αλλά να είναι μέλο τη ΤΟΑ ο τρίτο. have Και τώρα έχουμε πρόβλημα. Η Επιτροπή Ήτρε Βιομηχανίας ακόμα δεν έχει καλύψει τη θέση αυτή αλλά ακούω ότι θα είναι κάποιο Ισπανό σοσιαλιστή που είναι ταυτόχρονα και μέλο τη Επιτροπή Βιομηχανία και μέλο τη ΣΤΟΑ. Γιατί θα πρέπει να έχει και σχέση με την Επιτροπή Βιομηχανία και με τη ΣΤΟΑ. Καταλαβαίνετε τώρα που έχουμε βρεθεί, οι σοσιαλιστές διαμαρτυρήθηκαν ότι χτες αποφασίσαμε με λάθος προϋποθέσεις. Λοιπόν, θα ξαναπώ γερμανικά τώρα. Ε, αν ψηφίζαμε σύμφωνα με το σύστημα de Hunt θα ήταν σαφή τα πράγματα. Δεν μπορούν να πάνε τρεις σοσιαλιστές. Ένας μέχρι δύο, εντάξει. Το πρόβλημα είναι ότι αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα έχουμε μόνο τρεις σοσιαλιστές, θα έχουμε και τρεις Ισπανούς που θα πάνε στο Ναϊρόμπι. Έναν Ισπανό σοσιαλιστή από εμά αν ε, το δεχόμασταν αυτό που ψηφίσαμε, μια Ισπανίδα σοσιαλίστρια που είναι μέλος της βιομηχανία και της ΣΤΟΑ και έναν Ισπανό από το ΕΛΚ. Εγώ δεν έχω τίποτα κατά των Ισπανών. Αλλά αυτό το φόρουμ για τη διακυβέρνηση δεν είναι ε, τσιφλίκι των Ισπανών και πρέπει να προσέχουμε και αυτά τα πράγματα. Μίλησα σήμερα το πρωί με τον κύριο Ρόιλ ο οποίος έστειλε αυτή την επιστολή, δεν τη γνώριζε ε, την απόφαση του Προεδρείου και του είπα ότι χτες εμείς ε, ψηφίσαμε την κυρία Φερχόλ και του είπα να πει στους σοσιαλιστές ε, στην Επιτροπή Βιομηχανίας να ορίσουν την κυρία Μπαντία που είναι αναπληρώτρια στην Ήτρε. Οπότε έτσι με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Ε, είναι και θέμα των σοσιαλιστών να πείσουν τους ε, συναδέλφους τους ότι μπορεί να πάει σε αυτή τη θέση. Δεν είναι θέση της ΣΤΟΑ. Ενδεχομένως, πιθανώς, possibly, maybe. Εγώ δεν λέω possibly, εγώ αποφασίζω και ο κύριος Ρόιλ ότι δεν είναι possibly. Λοιπόν, ας αποφασίσουμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Αφού σας τα πω όλα αυτά, η κυρία Χάνιμπορ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι συνέβη, εμείς αποφασίσαμε χτες τις συνεδρίες των συντονιστών χωρίς να έχουμε τη γνώση αυτή. Γι' αυτό το επαναφέρω το θέμα. Νομίζω θα πρέπει να επανέλθουμε <laughs> στην απόφαση μας. Μέχρι στιγμής έχει ληφθεί μία απόφαση της Ήτρε που στέλνει ένα του ΕΛΚ. Γιατί στο Α δεν έχει ληφθεί απόφαση και η χτεσινή ψηφοφορία εδώ ήταν επί τη βάση ε, του γεγονότος ότι θα μπορούσε η κυρία Μπαντία να οριστεί από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Και άρα αποφασίσαμε να στείλουμε έναν του ΕΛΚ. Like because... Θα ήθελα να το ξαναδούμε παρακαλώ, διότι δεν είχαμε πλήρη γνώση των γεγονότων. Ε, και θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε. Επίσης ήθελα να πω ότι η κυρία Παντία έχει πολύτιμη εμπειρία σε αυτό το τομέα εδώ και καιρό και πραγματικά χρειάζεται μια συνέχεια εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Η πρόεδρος ε, εκτός ε, μικροφώνου. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξαναπούμε στις λεπτομέρειε. Είναι θαυμάσια η κυρία Πατία, είναι η σπουδαία, είναι η μεγαλύτερη, είναι τεράστια, είναι υπερδιπλάσια, αλλά... δεν θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία σε ένα νέο μέλος να κάνει τα ίδια όλα αυτά που έκανε η ίδια τόσο καιρό. Είναι και μέλο της Επιτροπής Βιομηχανίας αναπληρωματικό. Δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Μίλησα με το Ρόιλ και συμπιάστε τους δικούς σας στην Επιτροπή Βιομηχανίας να στείλουν την πατία είναι τόσο σπουδαία. Λοιπόν, η σκουρία σταμάτα εσύ. Εσύ μας έλειπε τώρα. <laughs> Όλοι γνωρίζουν πως έχει κατάσταση. Λοιπόν, α μείνουμε σε αυτό που είπαμε χθε. Ο κύριο Ρόιλ είναι πρόθυμο να το ξανακοιτάξει. Μίλησα μαζί του σήμερα το πρωί. Ε, είπε ε, ότι δεν ήξερα ότι πρέπει να στείλει κάποιο ψηστό. Η κυρία Χάνιμπολ, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένη. Μα ποτέ δεν είσαι, έχει το ανικανοποιητό αυτό. Ε, το πρόβλημά μου. Ναι, θα πρέπει να το ξαναψηφίσουμε όμως με βάση τόσο γνωρίζουμε σήμερα το πρωί που δεν ξέραμε χτε. Η πρόεδρο. Ωραία. Εάν δεν τηρήσουμε αυτό που ψηφίσαμε χτες, να ξαναψηφίσουμε. Θέλετε να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Μα δεν υπάρχει άλλη λύση, λέει η κυρία Χάνιμπολ, διότι η κατάσταση είναι καινούργια, έχουμε νέα δεδομένα. So, so, okay. You know the vote Γνωρίζετε ότι είναι πολύ απλή η ψηφοφορία. Ψηφίζουν οι συντονιστέ εκ μέρου των πολιτικών του ομάδων. Εντάξει, α ψηφίσουμε. Ο κύριο Κουρία. Γιατί είμαι υπέρ τη απόφαση που πήραμε χθε. Η κυρία Χάνιμπαλ, επόμενη, είναι υπέρ τη Μπαντία. Άλλη ομάδα. Liberate. please. Yesterday Εχθές και σήμερα Φερχάιν Ήτρε, ε, συμφωνούμε να τηρηθεί η χτεσινή ε, στάση μας, η χτεσινή πρότασή μας, μπαντία. Η συντηρητική, ούτε χτες το έκανα, ούτε σήμερα, δεν θα αλλάξω την ψήφο μου. Άλλος. Συντονιστής είναι παρόν, άλλη πολιτική ομάδα. Δεν είναι συντονίστρια δεν ξέρει τίποτα για την ψηφοφορία. Λήξει. Ψηφίστηκε η κυρία Φερχάιν. Κυρία Χάνι Μπάλμου, αν δεν το κάνετε εσεί, θα το κάνω εγώ. Θα πάω να πιάσω τον κύριο Ρόιλ. Του μίλησα και σήμερα το πρωί. Να πάρει ένα σοσιαλιστή. Πείστε τον. Βοηθήστε με. Εσεί είστε σοσιαλίστρια. Εγώ δεν είμαι και είμαι υπέρ τη Βαντία. Ελπίζω να είστε κι εσεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε τώρα εδώ. Ψηφοφορίες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τις κάρτες τις έχετε όλοι, έτσι. Δεν ξέρει κανείς, καμιά φορά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Κάβαντα Κύριε Καβαντά, θέλετε να παρέμβετε, να πάρετε τον λόγο. Παρακαλώ, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους που διευκόλυναν το έργο μας και μάλιστα σήμερα έχουμε και την εθνική αργία της Γαλλίας, εθνική ορτή, οπότε είναι διπλή η χαρά μας. Να τραγουδήσουμε τώρα το εθνικό σας ύμνο, τη Μασαλιότιδα ή όχι. Την επόμενη φορά θα έχουμε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για αλλαγή ύμνου. Τέλο πάντων. Λοιπόν, έχουμε 15 μέλη του ΕΛΚ, τρία παραπάνω από ό,τι κανονικά. Βερονίκ, εντάξει, οκ. So, the... Ξεκινάμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. 45 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 47 τροπολογία. Καταπίπτει. 47 δεν καταπίπτει, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 46 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 61 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Budget 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Γιούρι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Γιούρι 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 65 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Γιούρι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 68 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 69 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 71 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 67 αποσύρθηκε υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 83 υπέρ κατά αποχές ακαταπίπτει Καταπίπτουν όλες. Συγγνώμη, συγγνώμη. 85 ε, τώρα. Η 84, έτσι, υπέρ. 84 υπέρ, κατά και πάλι. Θα ήθελα να δω ποιοι ψηφίζουν υπέρ. 84 υπέρ, κατά, αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 84. Πέρας ψηφοφορίας. 7, 7 απορρίφθηκε. 85 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 86 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 88 και 89 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκαν 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 96 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 100 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 104 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 105 υπέρ κατά α, και πάλι 105 την ξέχασα πιο πριν, συγγνώμη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 106 την ψηφίσαμε. Ήδη 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ακαταπίπτει αυτή, συγγνώμη. Δικό σα φάλμα λέει η Πρόεδρος. Ωραία. Budget λοιπόν 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Γιούρι 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Γιούρι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 109 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 114 υπέρ κατά απόχέ. απορρίφθηκε 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 116 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 117 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 118 Budget 4 ε, γιατί αποσύρθηκε 118. 119 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Budget 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Budget 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 121-122 αποσύρθηκαν. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 125 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 127 αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε εντάξει. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 129 εδώ έχουμε παράτημα ναι, εντάξει υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 132 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 134 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 138 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η τροπολογία 144 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 1 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Recital A υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 και 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 11 αποσύρθηκε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 αποσύρθηκε 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Recital B υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Το C και D υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 16 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 18 και 19 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν Recital <coughs> C υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 20 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 21 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 24 αποσύρθηκε 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 26 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 29 υπέρ και 30 και 31 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Reciter A από την Επιτροπή Προπολογισμών υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 34, 35, 36, 37 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Recital και 38 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε recital D budget υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 41 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 43 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Recital B budget καλύπτεται από το ε δεν θα ψηφιστεί, εντάξει. Τελική ψήφος τώρα, ψήφιση με τις κάρτες σας. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε στην τελική ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. 23 υπέρ 2 εναντίον. Συγχαρητήρια κύριε Κάβαντα. Συγχαρητήρια θερμά. Ιδιαίτερα για 14η Ιουλίου, Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Μάλιστα. No, no, no, I'm not so bloody this morning. Δεν είμαι τόσο αιματοχαρή σήμερα, αιμοχαρή σήμερα το πρωί. no, but I, I, I, I... Yeah. During the war, huh? It goes very well with the Marseillaise. Huh? What do we do? No, we have. Nevedalova. Nevedalova. So, Κατερίνα, do you want to have... Κατερίνα, θες το λόγο. Είσαι εντάξει. Πάμε. Okay. Uh, very shortly, I would like to say... Θέλω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες τις από όλες τις πολιτικές ομάδες για την τόσο καλή δουλειά τους και ελπίζω να εγκριθεί. Ευχαριστώ. Πάμε, ψηφίζουμε. Okay. There are a lot of Μηπω uh, Μήπως καμιά φορά να ψηφίζουμε ε, συνδυασμένα μαζί, αν έχω αυτή την εντύπωση. Α, ένα, δύο, τρία μαζί. Ωραία. Ψήφι υπέρ. Δεν είστε. Ε, δεν θέλετε να τις ψηφίσουμε μαζί. Μπορείτε να καταψηφίσετε. Είστε υπέρ της υπερψήφισης των τριών αυτών ταυτόχρονα, όχι. Ένα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρι... Ε, απορρίπτεται. Δύο υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρία υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πέντε υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τι έγινε. Τέσσερα. Ξανά υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε, την ψηφίσαμε. Έτσι δεν είναι. Έξι, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εφτά υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμό ένα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μάρεκ γιατί δεν το ψηφίζουμε. Δεν πειράζει. 15. Α, 10 υπέρ. 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Έλεγχος χρειάζεται εδώ. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασα. 14 υπέρ, 11 κατά εγκρίνεται. Η 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τι λέει εδώ πήγαινε στην 28. 28 υπέρ, κατά. Ξανά, 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 Ορίστε. 23 τι έγινε. Μου είπαν να πάω στην 28. Έχει καταπέσει λέει εδώ. Έτσι δεν γράφει. 23 false. Και η 25 έχει αποσυρθεί. Πάμε στην 28. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 και 30 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά απόχέ. ε, απορρίπτεται. συμβασμό 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 36 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 40, όχι, μια στιγμή. Πάμε στην 39 και τη 40 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Και μία και η άλλη. Η 41 υπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 43 υπέ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 46 υπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό παρθών 4 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, Κατά. Έλεγχος. Αρχίζει ο έλεγχος για την 55. Πέρας. Accepted. Εγκρίνεται 18 υπέρ 6 κατά. Η 56 έχει αποσυρθεί. Και τώρα έχουμε εξτροπολογίες τη της Συμφωνείτε να τις ψηφίσουμε μαζί. Όχι. Υπέρ της 57. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κύριε Μιγκάλσκι, κατά αποχές εγκρίνεται. 60 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, τελική ψήφος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία και κλείνει μέσους. 23 υπέρ 2 κατά ευχαριστήρια κυρία Νεβέντ Αλόβα. Τώρα ψηφίζουμε το προϋπολογισμό, το περίφημο έγγραφο αυτό. Ο κύριος Λόκεγκαρτ θέλει και το λόγο. Πούντος, ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν. Τους σκιώδεις εισηγητές που ήταν πολύ καλοί συνεργάτες. Άκουσαν προσεκτικά τις απόψεις μεν των ΔΕ καθ' τη διάρκεια της διαδικασίας. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία και τους πολιτικούς μας συμβούλους για τον επαγγελματισμό τους. Τέλος, πολλές ευχαριστίες προς την Πρόεδρο, η οποία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ισχυρή και πυγμή για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Κατά την άποψή μου λοιπόν η Επιτροπή μα έχει σταθεί στο ύψο των περιστάσεων τροποποιώντα τον προπολογισμό αυτό και αποστέλλοντα ένα μήνυμα και προ την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι είναι στιγμή να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην εκπαίδευση και την νεολαία στον διαρκή αγώνα για να πετύχουμε την οικονομική ανάπτυξη και να βεβαιωθούμε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη για τον 21ο αιώνα στο διεθνέ προσκήνιο. Τα 45 εκατομμύρια για τη διαβίου μάθηση είναι ένα μεγάλο βήμα και το επόμενο σημαντικό βήμα είναι αυτό για τον αθλητισμό. Δείχνει ότι <clears throat> έχουμε μια ενοποιημένη προσέγγιση για το πρόγραμμα για τον αθλητισμό και τα απαραίτητα κονδύλια. Η Επιτροπή μας είναι ενωμένη στην προσπάθεια για διαφάνεια και ευθύ απαντήσεις ό,τι αφορά την επικοινωνιακή μα πολιτική και τα στρατηγικά σχέδια. Και ολοκληρώνοντα, να πω ότι χαίρομαι για το έργο που μας περιμένει τους ερχόμενους μήνες. Ιδιαίτερως γιατί η συνεργασία μας ως τώρα ήταν πολύ καλή σε πνεύμα αρμονικό. Ευχαριστώ όλους. Και σας πρόεδρε. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Λόκεγκάρτ. Δύσκολη η υπόθεση ήταν και πολλή δουλειά. Θα το καταλάβει κανείς αρκεί να κοιτάξει τα έγγραφα. Πάμε. Αρχίζουμε στην πρώτη σελίδα, καλό θα ήταν. Πρέπει να διαβάζω πάντα αυτά τα τρελά νούμερα εδώ πέρα. Ich Deutsch. Γερμανικά. 5.800 ψήφοι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5.801 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58.02 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58.03 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5805 υπέρ. Να λέω μόνο τα, τα τελευταία ψηφία. Το 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 06 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 07 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 08 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμό 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ α έχει αποσυρθεί 20 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, λανθάνουσα γλώσσα είπα πρώτα τα κατά Συμβιβασμός 2 ψήφι υπέρ ε, κρίνεται. 21 υπέρ. Α, όχι, όχι, όλα αυτά καταπίπτουν. Μέχρι το 29. Καλά, προχωράμε με ρυθμούς. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία για τη 30. Πέρας. 11-14 απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, τι έγινε, 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Λυπάμαι κυρία Μακλάκιν. Συμβασμός 3 ψήφι υπέρ κατά αποχές 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά ξανά ε, κατά αποχές εγκρίνεται τι λέει εδώ που πρέπει να πάω μα η 42 έχει καταπέσει το δικό σας έγγραφο ακολουθώ τώρα χάθηκα με μπερδέψατε με 44 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός Α. Τι είναι αυτό. Ε, για τα νούμερα του εισηγητή.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 Πρέπει να ψηφίσουμε για την εντολή του εισηγητή να αποκατασταθεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είμαστε σε διακοπέ και είναι θέμα ε, καταληκτική ημερομηνία. Ποιοι είναι υπέρ τη εντολή, ποιοι έχουν εμπιστοσύνη στον κύριο αυτό, υπέρ όλοι. Κατά κανεί. Ούτε και ο κύριο Νικάξη δεν είναι εναντίον. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Τι θα κάνουμε τώρα. Ms. Costa. Yeah. Yeah. I apologize, Lockegaard. Ζητώ συγγνώμη, Λόκεγκαντ. Ε, τέλειος η κυρία Τρούπελ, όπως και εκείνη πιο πριν. Πάντα δύσκολη δουλειά αυτή, η βρωμοδουλειά. Δεν βρίσκω τα χαρτιά. Πού είναι? Σίλβια Κώστα. Κώστα. I have a voting list I don't have. Give it to me. Βερονίκ, δώστε μου ένα πίνακα ψηφοφορία. Δεν έχω κατάλογο ψηφοφορία. Don't Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε τώρα. Αυτό είναι καβαδά. Όχι, Σίλβια Κώστα, εντάξει, πολύ καλά. Ξεκινάμε λοιπόν. Συμβιβασμός ένα. Η κυρία Κώστα πρώτα, συγγνώμη, η κυρία Κώστα. Απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις εξαιρετικές τους προτάσεις. Ελπίζω να είναι επικοδομητικό το αποτέλεσμα για όλους και κυρίως για την πλατφόρμα πολέμηση της φυλακής του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, συμβιβασμός ένα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 9 11 όχι 9 υπέρ 9 υπέρ κατά και πάλι 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Συμβασμό 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Συμβασμό 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 28 υπέρ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 απορρίφθηκε, απορρίφθηκε η 34. 35 υπέρ. Κατά. να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 35. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 17 υπέρ 8 εναντίον εγκρίθηκε. 36 υπέρ κατά και πάλι 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 40 υπέρ διαγραφή λέει για διαγραφή επί της ουσίας τροπολογία 40 υπέρ κατά απορρίφθηκε deleted 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 46 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τελική ψήφιση άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 23 υπέρ 2 εναντίον εγκρίθηκε συγχαρητήρια κυρία Σίλβια Κώστα so, Περνάμε τώρα στην έκθεση Τάκουλα, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού και τα λοιπά. Και τις άλλες να μου δώσετε παρακαλώ. Κύριε Τάκουλα, θέλετε να πείτε κάτι. Κοίταξε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη τους συνεργάτες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, τους σκιώδεις εισηγητές και ελπίζω ότι η ψηφοφορία ένα καλό αποτέλεσμα θα μας δώσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Περνάμε στην παράγραφα 1, τροπολογία 1 υπέ κατά, εγκρίθηκε συμβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 15 και 16 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν. Συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 24 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα 23 υπέρ δύο αποχές συγχαρητήρια κύριε Τάκουλα. So, nun zum Punkt 13. Και περνάμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Η ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό. Σαντιάγο, έχει τον λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια στιγμή, ένα δευτερόλεπτο, συγχωρήστε με, ψάχνω τα χαρτιά μου. Bueno, improviso igual, los tengo en inglés. <laughs> Sí. ε, <laughs> <clears throat> bien, ε... Λοιπόν, πολύ καλά. Ήδη είχαμε δύο ανταλλαγές απόψεων. Και σε αυτές νομίζω ότι ήδη είδαμε προς τα που πάει αυτή, ποια κατεύθυνση ακολουθεί η έκθεση. Πολλές ε, συναντήσεις είχαμε διάφορους ε, φορείς και σώματα και ενώσεις όσον αφορά τον βασικό αθλητισμό ερασιτεχνών και τους επαγγελματίες ε, αθλητές σε μια προσπάθεια συνθετική προσπάθησα να συνοψίσω σε περίληψη στον μικρό χώρο που έχουμε στη διάθεσή μας για εκθέσεις παρότι πιστεύω ότι με τη βοήθεια των πολλών σκιωδών εισηγητών και καθώς επίσης και με τους συντάκτες γνωμοδότησης των διαφορετικών επιτροπών μπορούμε να βελτιώσουμε βέβαια αυτή την έκθεση στο μέλλον. Θα ήθελα από την άλλη πλευρά απλά να σας διαβάσω το πρώτο σκεπτικό, την πρώτη αιτιολογική σκέψη, γιατί δείχνει κάπως την πορεία δηλαδή ο αθλητισμός συνεισφέρουν στην επίτευξη στατικών στόχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι έχει παιδαγωγικές αξίες και αρχές θεμελιώδεις και μπορεί να βοηθήσει στην ένταξη ε, των πολιτών άσχετα από φύλλο, εθνοτική προέλευση, υπηκότητα, κοινωνικό, κοινωνική κατάσταση, τάξη. Θέλω να τονίσω λοιπόν αυτήν την εγκάρσια ε, οριζόντια ε, ας το πω έτσι, μορφή του αθλητισμού ως χαρακτηριστικό. Και ακολουθώντας εκ του σύνεγγυ στην ανακοίνωση της ε, Επιτρόπου, νομίζω μια πολύ καλή ανακοίνωση είναι αυτή και έτσι επέτρεψε και σε σχέση με το άρθρο 155 ε, της Συνθήκης Λισαβόνας που όπως γνωρίζετε είναι η πρώτη φορά που δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασιστική δυνατότητα δηλαδή στην λήψη απόφασης για τα θέματα του αθλητισμού αρμοδιότητα να λαμβάνονται απόψεις για τα θέματα, ε, αποφάσεις για τα θέματα αθλητισμού για τα διάφορα κεφάλαια. Πρώτο, κοινωνική, ε, ε, κοινωνικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού. Τονίζουμε εδώ την προαγωγή, την προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία και στα αθλητικά κέντρα, ιδιαίτερα και όσον αφορά τα άτομα με ε, μειονεξίες, την καταπολέμηση κατά του ντόπινγκ. Ιδιαίτερα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διακίνηση των ουσιών αυτών για τον ντόπινγκ, καθώς επίσης και των ουσιών, ναρκωτικών ουσιών. Είναι ένα θέμα το οποίο μας ανησυχεί όλους και πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα για το μέλλον των αθλητών μας για να μπορούν να προετοιμάζονται και να προπονούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής όταν σταματάει η αθλητική τους δραστηριότητα. Ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι η απαγόρευση στα διάφορα στάδια για τους οπαδούς ή τους πιο βίαιους οπαδού δημιουργώντα ένα ευρωπαϊκό μητρό ώστε να απαγορεύεται η είσοδός τους στα στάδια στις κερκίδες ένα άλλο σημείο το οποίο αφορά και ε, τον αθλητισμό στο ευρωπαϊκό επίπεδο και το συζητήσαμε χθε με τον Πολωνό Υπουργό τη σπουδαιότητα που έχει ο αθλητισμό και όσον αφορά και τον αριθμό απασχολούμενων στον αθλητισμό γενικότερα και όσον αφορά και το ΑΕΠ στην Ευρώπη το οποίο συνεισφέρει. Αλλά θα ήθελα να τονίσω την ε, σπουδαιότητα του εθελοντισμού. Χωρί τον εθελοντισμό και τόσου πολλού εθελοντέ δεν θα ήταν δυνατόν να διασφαλίζουμε το αναβαθμισμένο αυτό επίπεδο στον αθλητισμό στην Ευρώπη. Κυρίως το ευρωπαϊκό επίπεδο αναβαθμίζεται με τις λέσχες και ομάδες ε, και μετά με τις ε, ενώσει, αθλητικές ενώσει, συλλόγους ε, κτλ. Υπάρχει και κάποιο άλλο σημείο το οποίο νομίζω είναι σημαντικό και αυτό είναι η καταπολέμηση. Ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πω η αναγνώριση της των χαρακτηριστικών των διαφορετικών ε, αθλητικών εκδηλώσεων. Αυτή η γνώση, αυτό το στοιχείο μπορεί να είναι σημαντικό. Μπορεί να είναι ένα στοιχείο καταπολέμησης των ε, στημένων παιχνιδιών, match fixing, καθώς επίσης ε, και της νόθευσης ε, των, ε, συναντήσεων. Είναι μια μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό. Τα αθλητικά, η άθληση πρέπει να μπορέσει να υποφελείται και από τα ταμεία, τα διαθετικά ταμεία και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι θα είναι πάντα ισχνά τα κονδύλια για τον αθλητισμό. Πρέπει να διασφαλίσουμε χρήματα, έτσι τα τα ταμεία θα μπορούσαν να δίνουν επιχορηγήσεις και στον αθλητισμό όπως γίνεται και για τον πολιτισμό και για άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Μετά στη συνέχεια ένα άλλο έχει επαναλαμβάνεται το ποιο είναι το ευρωπαϊκό αθλητικό πρότυπο. Είναι πολύ σημαντικό να το διατηρήσουμε και να το διασφαλίσουμε. Τονίζω την καλή διακυβέρνηση και διαχείριση στον αθλητισμό που βασίζεται κυρίως πρέπει να βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και δημοκρατικότητας και όλα τα συμβαλόμενα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να εκπροσωπούνται επαρκώς στα αθλητικά όργανα που ε, συμμετέχουν στους διάφορους φορείς. Επίσης τη σπουδαιότητα, τη σημασία του να δεχτούμε, του να υπάρχουν αντισταθμίσεις όσον αφορά τους παίκτες. Αυτό είναι σημαντική υποστήριξη για τις λέσχες. Ζητούμε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μητρώου για τους φορείς εκείνους όπου θα αναφέρεται, θα αναφέρονται από πλευρά τους ποιοι είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν αυτούς που τους εκπροσωπούν, ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος. Ε, χρηματοοικονομική δικαιοσύνη. Ο κύριος Ντεάν αυτή τη στιγμή συντάξει μια σημαντική έκθεση για την ε, χρηματοοικονομική διαφάνεια των οικονομικών, των συλλόγων και ομάδων. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Και ένα άλλο σημείο το οποίο συζητήθηκε σε σχέση με την Πολωνική Προεδρία είναι η διασφάλιση του ακέραιου χαρακτήρα, έντιμου χαρακτήρα των εκδηλώσεων. Πρέπει να υπάρχει ποινική νομοθεσία για κυρώσει στην Ευρώπη με παρόμοιο τρόπο, συγκρίσιμο τρόπο, ώστε να υπάρχει κύρωση αυτού του αδικήματο όταν νοθεύονται οι εκδηλώσει, οι αθλητικέ συναντήσει. Καθώ επίση ε, και σε σχέση με την ύπαρξη ε, κάποιου φορέα που θα μπορούσε να επιλαμβάνεται των δικαστικών, δικονομικών αυτών θεμάτων είτε στι Βρυξέλλε ε, για παράδειγμα ε, λόγω του κοινοτικού δικαίου υπάρχει ε, μια, αντιπροσωπία μια ε, δυνατότητα τέτοια αντιπροσωπία για τις είπα και για την Αυστραλία γιατί να μην έχουμε κάτι τέτοιο και εμείς οι ίδιοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες, ένα άλλο κεφάλαιο, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι πολλές φορές συμβαίνουν τέτοιου είδους γεγονότα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στημένα παιχνίδια, στοιχήματα, όταν λαμβάνονται συμφωνίες με αυτές τις χώρες πρέπει να λαμβάνονται και υπόψη και αυτά τα θέματα. Και επίση να ζητήσουμε από τι λέσχε και ομάδε να εποπτεύουν τα θέματα των ανηλίκων. Να είναι υπεύθυνοι όταν για παράδειγμα ε, προσλαμβάνεται κάποιο ανήλικο σε κάποια ομάδα η λέσχη να μην παραμένει μετά ασυνόδευτο ή ε, χωρί φροντίδα αλλά να μπορεί να ε, τον φροντίζουν και να την χάνει μέρημνα. Ένα άλλο πρέπει να είναι ο Ευρωπαϊκό Φορέα για τον Αθλητισμό. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα να διοργανωθεί μια Ευρωπαϊκή ημέρα για τον αθλητισμό, όπως έχουμε μια ημέρα για τόσα άλλα πράγματα, ώστε σε κάθε πόλη, σε κάθε χώρα να μπορούν να αποφασίζουν το τι θα γίνεται, αλλά θα είναι μια μέρα που θα είναι αφιερωμένη στο αθλητισμό ώστε και να έχουμε και τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής πρωτεύουσα αθλητισμού με υποστήριξη, με επιχορήγηση ή άλλη ε, δυνατότητα συνδρομής. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Αθλητικών Δραστηριοτήτων ε, γηγενών αθλητικών δραστηριοτήτων. Ενδιαφέρον θα ήταν να είχαμε ένα φεστιβάλ επίδειξης αυτών των γηγενών αθλητικών δραστηριοτήτων από πλευράς κάθε χώρα χώρας και ε, ένα πρόγραμμα για νέους αθλητές τύπου Έρασμος. Γνωρίζουμε ότι βρίσκεται κάτι του υπομελέτη αλλά να συμπεριληφθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο και θα ήθελα να αποκαταστήσω, να καταστήσω σαφές το ένα ή άλλο θέμα διότι από πλευράς ε, ε, του Βρετανικού τύπου είχε αναφερθεί αυτό το θέμα χωρίς να γνωρίζουν όμως την ουσία του θέματος. Υποβάλλω μια πρόταση ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Σημαία να συνοδεύει ε, στον, ε, στα διάφορα στάδια της εκδηλώσεις. Είναι ανοιχτό αυτό προς έγκριση ή μη και στις διάφορες ε, εκδηλώσεις όταν συναγωνίζονται, ανταγωνίζονται οι διάφοροι αθλητές μπορεί να έχουν το εθνόσημό τους αλλά επίσης να έχουν και την ευρωπαϊκή σημαία, το ευρωπαϊκό σύμβολο. Αυτό όμως δεν θα είναι υποχρέωση. Κάθε χώρα, κάθε αντιπροσωπεία θα αποφασίζει αν αυτό είναι αποδεκτό και σκόπιμο ή όχι θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για όλη την υποστήριξη που μου έδωσε για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης και επίσης φυσικά είναι αυτονόητο για όλου όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου στους κόλπου του ΕΛΚ και στο ίδιο το γραφείο μου Γνωρίζετε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα και αισθάνθηκα πραγματική υποστήριξη, αυθεντικά ομόφωνη υποστήριξη, ομόθυμη υποστήριξη υπέρ του αθλητισμού. Είναι η πρώτη έκθεση αυτή. Προσδοκώ αδειμονώ να ακούσω τις, τα σχόλιά σας και τις τροπολογίες που θα υπάρξουν και έτσι να μπορέσουμε με τη γραμματεία να ε, επεκτείνουμε κάπως την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Μου είχαν πει τέλη Αυγούστου θα κλείσει, αλλά θα είμαστε σε διακοπές ούτως ή άλλως τότε. Και γι' αυτό για να διευκολύνουμε να μπορέσουν να κατατεθούν αυτές οι τροπολογίες Ίσως να μπορέσουμε να επεκτείνουμε κατά μια εβδομάδα την ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών, την καταληκτική ημερομηνία για να βελτιωθεί η έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και αναμένω και προσδοκώ στα σχόλιά σας. Α, θα τα πάρετε τα σχόλια μου αγαπητοί ε, κύριε. Εισηγητά. Ε, και ε, αυτοί που γελάτε θα τα συζητήσουμε, θα τα ξαναπούμε τα θέματα της Ευρωπαϊκής Σημαίας. Ναι, ναι, Λοιπόν, κύριε Κέλλη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για τα πρακτικά. Δεν είναι επίκριση, τίποτα τέτοιο. Αλλά δεν μπόρεσα να ψηφίσω σήμερα το πρωί, δεν κατάλαβα γιατί. Το δέχομαι γιατί ισχύει και για άλλους, αλλά το σύστημα χρειάζεται να το ξανακοιτάξουμε από πλευράς κοινοβουλευτικής. Δεν έχει να κάνει με την Επιτροπή Πολιτισμού. Υπάρχουν μέλη τακτικά, αναπληρωματικά που συμμετέχουν στι συζητήσεις κτλ. Και δεν μπορούν να ψηφίσουν ούτε τι δικέ του τροπολογίε ή τι τροπολογίες που έχουν επεξεργαστεί το σύστημα να ξανακοιτάξουμε αυτό προ το παρόν. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να ψηφίσω και αφού ε, δεν μπορούσα να ψηφίσω μελέτησα την έκθεση του κυρίου Φίσα. Ε, χαίρομαι γι' αυτό. Πρέπει να σα πω ότι είναι εξαιρετική. Καλύπτει όλες τις βασικές διαστάσεις που πρέπει να καλύψουμε και τονίζει που χρειάζεται δράση εν ευθέτω χρόνο. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φίσας για την καταπληκτική του δουλειά. Μερικά σημεία που χρειάζεται και αξίζει να επαναλάβουμε. Μίλησε για τις αθλήτριες. Οι γυναίκες στον αθλητισμό είναι ένα θέμα που είναι σοβαρό, ε, που είναι διαρκές και ένα από το θέμα γιατί δεν έχουμε τόση συμμετοχή και τόση αναγνώριση των γυναικών στον αθλητισμό είναι διότι δεν εκπροσωπούνται στα υψηλά επίπεδα ε, των αθλητικών ε, οργανώσεων και ηγεσιών. Το είπε και ο ίδιος ο ηγητής, έχει δίκιο. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε και πάλι την οικονομική αξία του αθλητισμού. Πολλοί που δεν ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό δεν το αναγνωρίζουν. 6,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ είναι. Είναι τεράστιο. Και επίσης υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό για να απτυχθεί ο τουρισμός ως κλάδος της οικονομίας. Και οι εθελοντές είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το τονίζει και ο συγητής. Και επίσης αναφέρει και κάτι άλλο που είναι ένα μόνιμο πρόβλημα για τον αθλητισμό. Είναι η σύγκρουση των εθνικών ομάδων με κάποιους αθλητικούς συλλόγους. Και θα πρέπει να αναγνωριστεί ε, ότι θα πρέπει ε, αθλητές να αφήνονται ελεύθεροι όταν τους χρειάζονται οι εθνικές ομάδες και να μην τους δεσμεύουν οι σύλλογοι στους οποίους αγωνίζονται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η σωστή χρηματοδότηση του αθλητισμού είναι επίση πολύ σωστό. Για τα διαρθρωτικά τιμία θέλω να μιλήσω. Έχω κάνει και ε, τροπολογία ψηφίστηκε, εγκρίθηκε και ανοίγονται τώρα νέε δυνατότητε για τη χρηματοδότηση και από τα διαρθρωτικά ταμεία. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τους managers, τους ε, προσώπους των παικτών, θα πρέπει να το δούμε αυτό και το αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο για να επιλύει διαφορές και προβλήματα ε, που δεν μπορούν να λυθούν σε εθνικό επίπεδο. Θα Μα απαλλάξει από πολλούς μπελάδε να υπάρχει ένα τέτοιο δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, μιλάει για την Ευρωπαϊκή Μέρα του Αθλητισμού και για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Αθλητισμού. Βεβαίω, να έχουμε μια πολιτιστική πρωτεύουσα αθλητισμού στην Ευρώπη και όσο για την Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητισμού να γίνονται ακριβώς εκείνη τη μέρα εκδηλώσεις στι εκάστοτε πολιτιστικέ πρωτεύουσε, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα τα χωριά και όλες τις πόλεις αλλά στις πρωτεύουσε, ε, τις πολιτιστικές θα μπορούσαμε να το κάνουμε και για τη σημαία γιατί όχι, γιατί να μην κυματίζει τις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις γιατί υπάρχει κόσμος που δεν τη σκέφτεται καν τη σημαία δεν του περνάει από το μυαλό μόνο η εθνική του Καλό θα ήταν να έχουμε και την Ευρωπαϊκή Σημαία, θα μας φέρει πιο κοντά στους πολίτες και στον αθλητισμό τους πολίτες. Γίνεται λόγος και για γηγενή αθλήματα και είδη ε, αγωνισμάτων. Έχουμε ένα χάρτη, είπε ότι ορισμένα έχουν εξαφανιστεί, ε, έχουν εκλείψει. Καλό θα είναι να έχουμε ένα τέτοιο χάρτη να συγκεντρώσουμε γιατί είναι και θέμα πολιτιστικής ποικιλομορφίας και στον αθλητισμό στην Ευρώπη. Είναι πολύ καλή έκθεση λοιπόν και συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Ε, και συμφωνώ ίσως να παραταθεί η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες γιατί τέλη Αυγούστου θα είμαστε όντως σε διακοπές ή αν όχι σε διακοπές θα είμαστε σε διάθεση διακοπών και δεν θα κάνουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Για την πρώτη σας παρέμβαση θα ήθελα να επανέλθω. Έχετε κάθε δικαίωμα να υποβάλλετε τροπολογίες, να ομιλείτε. Είστε από τους πιο επιμελείς συναδέλφους εδώ. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είστε αναπληρωματικό μέλος. Γι' αυτό μπορείτε να ψηφίσετε μόνο όταν απουσιάζει τακτικό. Ε, όταν είναι δική σας τροπολογία να συμφωνήσετε με κάποιο συνάδελφο να ψηφίσετε στη θέση του. Αλλά είναι υπέρ της τροπολογίας σας έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες γιατί εσείς είστε ένας τόσο επιμελής αναπληρωματικός. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά να το λύνουμε μεταξύ μας. Εντάξει, ας τα αφήσουμε εδώ κύριε Κέλλη. Εντάξει, σύντομα σας παρακαλώ. Συγγνώμη. Ναι, ναι, απολύτως. Δεν το κάνω ζήτημα εγώ προσωπικό, απλώς σας λέω ότι πρέπει να το κοιτάξουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί, ε, να το κοιτάξουμε αυτό στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Εντάξει, ε, λειτουργεί όπω όλα τα άλλα κοινοβούλια. Υπάρχουν τακτικά μέλη που ψηφίζουν και αναπληρωτέ ψηφίζουν ε, όταν λείπουν οι τακτικοί γιατί είναι στον πάγκο. Παντού σε όλα τα κοινοβούλια. Λοιπόν, 13 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θέλετε να πάτε και σπίτια σας σήμερα. Θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε και να μην πείτε όλοι αυτά που είπαν οι προλαλήσαντε. Εντάξει. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι και μην αρχίσετε μια φορά και ένα καιρό, Αδάμ και η Εύα, τα ξέρουμε αυτά. Η κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Φίσας, και εσείς ε, χτες ε, είπατε πολλά. Ε, ε, λίγα έχουμε να προσθέσουμε με τροπολογίες και θα κάνω προ... τροπολογίες και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και σε επίπεδο ε, Επιτροπής ε, Ελευθεριών που προετοιμάζω τη γνωμοδότηση εγώ. Καμιά φορά όταν κάνουμε τις συζητήσεις υπάρχει κίνδυνος να κυριαρχεί το ποδόσφαιρο. Καθόλου όμως στην έκθεσή σας δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις σύντομες Κάτι που μου λείπει, όχι από την έκθεσή σας, από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι οι δράσεις. Πού είναι οι δράσεις. Να δούμε, ε, να το προτείνουμε εμείς στην έκθεσή μας, εφόσον δεν το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον ντόπινγκ, ας πούμε. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν θα πρέπει να πέσουν θύματα ε, στην καταπολέμηση ε, ε, του ντόπινγκ. Βεβαίως ο καθαρός αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά έχουν και δικαίωμα σε μια ιδιωτική ζωή οι αθλητές. Σε ό,τι αφορά τη διπλή καριέρα, dual career, είναι σημαντικό, το έχω συζητήσει και με πολλούς αθλητές. Μέχρι το γυμνάσιο καλά τα πάνε, αλλά μετά το γυμνάσιο δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα για να μπουν στο πανεπιστήμιο ή να έχουν ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση ε, ειδικά όταν είσαι αθλητής που αλλάζει συχνά συλλόγου, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις και σπουδές ταυτόχρονα. Και... Όμως είναι σημαντικό να έχουν και δίπλωμα ε, οι αθλητές πανεπιστημιακό σε ό,τι αφορά το διαιτητικό δικαστήριο είπε και ο υπουργό ε, θα μπορεί να προσφεύγει και ο κόσμος, οι πολίτες εκεί. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώ εννοείται με το αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο. Για τους μάνατζερ, τους εκπροσώπους των παικτών, ναι, συμφωνώ με το Μητρό. Αυτά που προβλέπει η FIFA δεν είναι αρκετά. Και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, υπάρχει και το μπάσκετ και το ράγμπι και δεν υπάρχει το σύστημα TMS στα άλλα αθλήματα παρά μόνο στο ποδόσφαιρο. Και αυτό χρειάζεται να το κοιτάξουμε. Αυτά. Και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μιγκάλσκι. Σας ευχαριστώ λίγο περισσότερο κριτικό πνεύμα. Φοβούμε ταυτόχρονα ότι η έκθεση θα κάνει τον κόσμο να αντιπαθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να την συμπαθήσει. Διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί σε ο πλαίσιο τη έκθεση. Θα επισημάνω τρία-τέσσερα τέτοια πραγματάκια που νομίζω ότι δεν είναι σωστό ότι εντάχθηκαν σε αυτό το πλαίσιο τη έκθεση. Υπάρχει αρχή ότι δεν θα πρέπει να δημιουργείται κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαίο πρώτα απ' όλα. Πολλά τα πράγματα έχετε πιστεύω εντάξει στο κείμενο. Στο ε, ναι, τι αναφέρεται. Τονίζετε εκεί και λέτε πόσο σημαντική είναι η μεταφορά δικαιωμάτων με βάση ένα πρότυπο το οποίο θα ήταν κεντρικού σχεδιασμού. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς ε, περί τίνος πρόκειται εδώ μπορεί κανείς να υποθέσει ότι θα έχει αρνητική έκβαση στο τέλος. Επίσης προτείνεται ένα ευρωπαϊκό μητρό ε, ατζέντιδων ή πρακτόρων των παικτών ή των αθλητών και αυτό φαίνεται να είναι περίτω. Θέλετε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό φόρουμ για την διαιτησία και αυτό είναι δαπανηρό επιπλέον. Θα έπρεπε να ζητηθεί από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους αν θεωρούν ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία τα έσοδα τα οποία προέρχονται από τους φόρους τους που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Επίσης αναφέρεται μία ημέρα για τον αθλητισμό. Έχετε δίκιο σε σχέση με την ε, ε, ημέρα που υπάρχει ήδη. Χρειάζεται μια δεύτερη για να ε, γιορτάζουμε τον αθλητισμό. Επίσης προτείνεται πρωτοβουλίες για μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα αθλητισμού Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού. Δεν θα έχει νόημα να δημιουργηθεί και άλλη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτιστική για τον αθλητισμό και για το 26 ενδιαφέρον σε σχέση με το βρετανικό τύπο αλλά επίσης ευρύτερα σχολιάστηκε και στον τύπο στην Πολωνία πρέπει να σας πω Πρόκειται για ευρωπαϊκές εκδηλώσεις όπου η ευρωπαϊκή σημαία θα έπρεπε να τις συνοδεύει. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο, στα ρούχα και στον εξοπλισμό των αθλητισμών θα πρέπει να υπάρχει το σύμβολο αυτής της ευρωπαϊκής σημαίας. Αξιοπερίεργο πρέπει να πω αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Αν το εθνικό σύμβολο της Πολωνίας είναι ο αετός, τι προτείνεται. Τα ευρωπαϊκά στεράκια της ευρωπαϊκής σημαίας να αντικαταστήσουν, να υποκαταστήσουν τον Αϊτό, να πάνε γύρω από τον Αϊτό. Πώς τεχνικά βλέπετε μια τέτοια δυνατότητα και ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος μιας τέτοιας πρότασης. Ευχαριστώ. Uh, hello. <coughs> Uh, okay. Uh, well, I'd like to start by... Να ξεκινήσω λέγοντας ότι σε όσα είπε ο κύριος Φίσερ έχει αρκετό δίκιο η ισοτιμία είναι κάτι που το εμπνέει ο αθλητισμός και εγώ έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο σε όλες τις κατηγορίες. Δίνουν, δίνουν τα αθλήματα φιλοδοξίες και ελπίδες στους ανθρώπους, φέρνουν πιο κοντά τις κοινωνίες, ανθρώπους από διαφορετικές θρησκείες, κοινωνικές τάξεις, τους φέρνουν πιο κοντά. Είναι πολύ λοιπόν λογικά πολλά από αυτά που προτείνει. Όμως για το 26 Πρέπει να πω ότι όταν το διάβασα δεν ήξερα να θέλω να κλάψω ή να γελάσω. Διότι δείτε τι λέει σήμερα εδώ η εφημερίδα. Είναι η ίδια σημαία που προτείνουμε. Κοιτάξτε, η Daily Express είναι. Το Όχι καμία του Μέρντοχ. Μιλάμε για την ίδια σημαία που λέτε και στα ρούχα των αθλητών να υπάρχει και στι μεγάλε αθλητικέ εκδηλώσει, αλλά δεν έχει δεχτεί το Σύνταγμα. Δεν έχει γίνει τόσο δεκτή. Άρα δεν ξέρω πόσο δημοφιλή θα σε όλη την Ήπειρο. Πρόσφατα σε δημοσκόπηση στο Ηνωμένο Βασίλειο φάνηκε ότι το 50% τουλάχιστον θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κοιτάξτε τι θα γίνει αν σε μεγάλε αθλητικέ εκδηλώσει σχηματίζει αυτή η σημαία ο Πίτερσον, ο Βίλκινσον θα θέλουν να φοράνε στις στολές τους τη σημαία. Νομίζω ότι θα είναι... Δεν θα είναι καθόλου θετικό. Ορίστε, έχετε τηλεοράσεις, εφημερίδες, ό,τι τι άλλο θέλετε. Και κάμερα σας τραβάει, μια χαρά είστε. Ευχαριστώ. Μα δεν με συζητάμε για τέτοια μικροπράγματα. Πολιτική κάνουμε εδώ και καλή. Και το θέμα της σημαία είναι πρόταση. Ακούσαμε. Να διαβάσετε. Είναι πρόταση. Προτείνει. Δεν είναι υποχρέωση. Και ο Βρετανικός τύπος νομίζω αφήστε καλύτερα. Εντάξει, α μην το συζητήσουμε. Ο κύριος Μπελέτ. Thanks very much, uh, Chairman. Uh, στα αγγλικά κύριο Μπελέτε. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα ω σκιώδη εισηγητή, να πω ότι μια τροπολογία θα την υποβάλω ώστε να ζητήσω η σημαία του Μέρντοκ να υπάρχει σε όλα στις ελληνικές εκδηλώσει και στον Βρετανικό τύπο. Ίσως να είναι καλύτερη για ευρωπαϊκή σημαία και να μας εξυπηρετήσει αυτό. Τέλος πάντων συγχαρητήρια στον εισηγητή ο οποίος και φιλόδοξο είναι και ρεαλιστικός στις προτάσει του. Σαντιάγκο τα μέσα μαζική ενημέρωση ε, δεν ήταν περίεργο που ξεκίνησαν τα φιλικά πειρά. Όμω αυτό που με εκπλήσει είναι ότι πολλοί συνάδελφοι παρεμήνευσαν και παρανόησαν πολλέ από τι προτάσει τη πρόταση. Όταν λέμε για, την, για τον σταθμό του Αθλητικού Δικαστηρίου. Δεν προτείνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να τον αναλάβει αυτό. Είναι κάτι που αποτελεί αυτοδιαχείριση, αυτοδιακυβέρνηση. Δηλαδή οι φορεί, τα σώματα που είναι υπεύθυνα να αναλάβουν την ευθύνη. Δεν λέμε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί θέλουμε καλή διακυβέρνηση και στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα. Δεν θα ήθελα να λάβει όμω την πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' αυτή. Το ίδιο και για άλλε προτάσει. Για παράδειγμα, για τους για τις ενώσεις των αθλητών, όταν λέμε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγραφής. Δεν λέει οι συνάδελφοι, οι συγκεντές να οργανωθούν αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε να στηριχθεί, να στηριχθούν οι Διαπραγματεύσει που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα μεταξύ των μάνατζερ, των ε, ενώσεων των παικτών και, των, ε, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι εμείς να αναλάβουμε τη διοργάνωση. Δεν το λέει αυτό η έκθεση και μην τα πείτε αυτά και στο Βρετανικό τύπο. Διότι είναι ανοησίες και ψέματα αυτά. Και να ολοκληρώσω με δύο πρόσθετες παρατηρήσεις, Πρόεδρε σε κάτι που αναφέρει ο εισηγητής, πολέμηση της διαφθοράς, καταπολέμηση της, ε, των στημένων παιχνιδιών. Εδώ λοιπόν ε, για τις οικονομικές αυτές ε, παρεκκλήσεις πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις και να πάρω και ένα παράδειγμα από τη Λίγκα, την Ευρωλίγκα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε ένα παράδειγμα με την πρώτη εθνική της Αγγλίας στη Μάντσεστερ, όπου 400 εκατομμύρια αγγλικές λίρες ε, ήταν το εισόδημα από τα διαφημιστικά σποτ. Η ευθεία των σπόνσορας μόνο αποκόμισε τόσα. Άρα οι αιτήσει μας για διαφάνεια, για να δούμε πώς λειτουργούν οι σπόνσορε, είναι σημαντικό για να υπάρχει ισοτιμία στους κανόνε. Μιλάμε για ευρωπαϊκούς αγώνες, για, για ευρωπαϊκό συναγωνισμό, για την UEFA, για να υπάρχει ένα σύστημα με ίσους κανόνες. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση, η οποία είναι αυτοδιακυβέρνηση. Θέλω να πω στον συνάδελφο που δεν είναι μέλο αυτή τη κοινοβουλευτική επιτροπή, καλό είναι ότι συμμετέχετε σήμερα. Θέλω να σα πω ότι στη συνθήκη αναφέρεται ότι οι αθλητικέ ενώσει και σύλλογοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, να έχουν την αυτονομία του. Κανένα από εμά δεν θέλει να αναμειχθεί σε αυτά. Αν κάποιο από την FIFA, από την UEFA ή από άλλε ενώσει ή συλλόγου ζητηθεί να βοηθήσει κάτι, ώστε να υπάρξουν κανόνες και κανονισμοί και ρυθμίσεις, τότε θα πρέπει να βοηθήσουμε να τηρηθεί αυτό. Δεν το κάνουμε εμείς. Μια πλατφόρμα θέλουμε να βοηθήσουμε να εξευρεθεί. Είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα από αυτό που διαβάζετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσείς διαβάζετε κάτι και του δίνετε ερμηνεία που δεν εμπεριέχεται στο κείμενο. Ο κύριος Μόρης παρακαλώ. Και εγώ θα μπορούσα να μιλήσω για τη σημαία, αλλά δεν ήθελα αυτό να ε, μας κάνει να παραμελήσουμε τα άλλα σημεία αυτής της πολύ καλής έκθεσης. Για... Όσο σε πω λοιπόν. Είναι μια έκθεση που την περιμέναμε καιρό, ιδίως στον αθλητικό κόσμο της Ευρώπης. Είναι αρκετά πλήρης, ιδίως μετά τις δηλώσεις του Υπουργού για τον αθλητισμό, του Υπουργού της Πολωνίας για τον αθλητισμό. Μπορώ να πω ότι όσα αναφέρει η έκθεση θα φροντίσουμε να προωθηθούν το ερχόμενο εξάμεινο. Η συνδίκη τη Λισαβόνα μα επιτρέπει να διαθετήσουμε τη δραστηριότητά μα και σε αυτόν τον τομέα. Άρα, να στηρίξω τον συνάδελφο Φίσα και να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το σύστημα διαφάνεια των ίσων κανόνων του fair play στο, στον αθλητισμό είναι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των μελλοντικών, των επόμενων γενιών. Επίσης θέλουμε να υπάρχει και μια προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς να δούμε κατά πόσον υπάρχει ένα σύστημα για όσους, ε, μάλλον να καταπολεμήσουμε το σύστημα που επιτρέπει να ανθεί η διαφθορά. Και επίσης η σημαία νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει αντίφαση. Δεν υπάρχει θέμα με το γεγονός ότι εγώ είμαι Πολωνός, ο κύριος Φίσας Ισπανός, η πρόεδρος Γερμανίδα. Τι πρόβλημα υπάρχει. Γιατί να υπάρχει αντιπαράθεση. Μιλάμε για ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το 2012 λοιπόν, εάν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα οι Γερμανοί και οι Πολωνοί αθλητές βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό, μπορούν να βλέπουν να κυματίζει γύρω τους η εθνική του σημαία και η ευρωπαϊκή. Είναι σημαντικό αυτό για τους πολίτες όλους και νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να το στηρίξουμε. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιοι τομεί, όπω ο αθλητισμό, που έχουν μια σημαντική εθνική αλλά και διεθνή διάσταση. Και αυτό είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Είναι δύσκολο να βρούμε κάτι ανάλογο. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι η αρχή τη επικουρικότητα εδώ θα εφαρμοστεί για να μην πιέσουμε τα πράγματα άναθεν και επιβάλλουμε αποφάσει. Για τον αθλητισμό, λοιπόν, για πρώτη φορά πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε του αθλητέ στην Ευρώπη. Όχι οι αθλητέ να μα βοηθήσουν να οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια σειρά παραδειγμάτων στην έκθεση που δείχνει ότι ε, επικεντρωνόμαστε στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αλλά δεν κοιτάζουμε να βοηθήσουμε τον αθλητισμό αυτό καθεαυτό. Η πρόταση είναι να υπάρχει ευρωπαϊκή σημαία σε εθνική και συναντήσει Είναι κάτι τελείω παράλογο ας πούμε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μα έχει τεράστιο ρόλο το ποδόσφαιρο λόγω χάρη για την εθνική μα ταυτότητα, την εθνική μα ε, ε, ιστορία. Η Ουαλία και η Σκότια δεν έχουν την ε, σημαία της Αγγλίας στα κήπεδά του, Άρα είναι πολύ σημαντικό για μα. Είμαστε παθιασμένοι, έχουμε μεγάλη, μεγάλο ενθουσιασμό για τι εθνικέ μα ομάδε. Εδώ προτείνεται ευρωπαϊκή ταυτότητα, αλλά δεν μπορεί κανείς να την επιβάλλει στους ανθρώπους και στους φιλάθλους. Εάν επιμείνουμε σε αυτό, νομίζω ότι θα απομακρύνουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το πώς, ε, διαιτητικό δικαστήριο και το πώς αυτό θα επηρεάσει εάν υπάρχει ένα θέμα μεταξύ ενός, ε, μιας πλευράς ευρωπαϊκής και αν η άλλη πλευρά είναι εκτός Ευρώπης. Μπορεί να προκύψουν δυσκολίες. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πώ αντιμετωπίζουμε τον αθλητισμό. Διότι τα περισσότερα από τα σχόλιά μα φαίνεται να αφορούν ιδίω το ποδόσφαιρο. Δείτε τι γίνεται σήμερα και σκεφτείτε τι θα γίνει στην διάσταση, για τη διάσταση του αθλητισμού στο μέλλον. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που επικεντρωνόμαστε στην εκπαίδευση και στο τοπικό επίπεδο για του παίκτε και του αθλητέ, αλλά υπάρχει και η διάσταση τη κοινωνική συμπερίληψη. Ε, η δύναμη του αθλητισμού να φέρνει του ανθρώπου κοντά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε και όχι πώ θα διαμορφώσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα στον αθλητισμό. Λοιπόν, το λέω τώρα, άπαξ διαπαντό. Η έκθεση αυτή δεν είναι έκθεση για την ευρωπαϊκή σημαία. Η έκθεση αυτή δεν ε, ε, εντάσσει και πουθενά αλλού τη σημαία. Είναι μια φανταστική έκθεση για πάρα πολλά σημαντικά θέματα στον αθλητισμό. Έχει και μια πάρα πολύ μικρή πρόταση. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα όσοι πάρετε το λόγο δεν χρειάζεται να εξηγήσετε γιατί δεν ισχύει αυτό. Μπορεί και να μην περάσει. Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει την πρόταση. Μια φρασούλα είναι σε αυτή τη θαυμάσια έκθεση. Και αν δεν έχετε να πείτε τίποτα άλλο παρά για τη σημαία, ε, τότε καήκαμε η Επιτροπή μας θα πρέπει να προτείνει περισσότερα πράγματα από μια σημαία απλούστατα. Γελιοποιούμαστε. Εάν επικεντρωνόμαστε σε αυτή τη μικρή προτασούλα, αυτά, τίποτα άλλο. Α είμαστε λίγο πιο σοβαροί, γιατί η έκθεση είναι σοβαρή και καλή και σπουδαία και λέει και σημαντικά πράγματα. Τώρα μην ακούσω καρά για τη σημαία. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση. Φυσικά είναι πολύ ενδιαφέρον να γίνεται λόγος ε, για τους αθλητές και για την ίδια κοινωνική ασφάλιση για αυτούς, όπως και για τους εργαζόμενους. Πολύ συχνά συμβαίνουν ατυχήματα στα αθλήματα και θα πρέπει να καλύπτονται οι αθλητές. Πολλές φορές δεν έχουν και άλλα επαγγέλματα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πτυχή της ασφάλισης έναντι ατυχημάτων των αθλητών για, ελπίζω ότι η Επιτροπή, από την Επιτροπή θα θέλαμε να ακούσουμε ποια πρόταση ε, θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και για τα διαθροτικά ταμεία, για τη βοήθεια εκεί όπου μπορεί να υπάρξει υποστήριξη είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρονται και οι ενώσεις και σύλλογοι ερασιτεχνών αθλητών, δηλαδή μη επαγγελματιών, καθώς επίσης και κινητικότητα ή προγράμματα κινητικότητας για τους αθλητές. Ελπίζω να μην υπάρχει εδώ, να μην είναι θέμα μεταφραστικού σφάλματος. Δεν θα έπρεπε να αναφέρεται αθλητές, αλλά νέοι, νέοι, αθλη, ε, ε, Ίσως θα μπορούσε αυτή η μικρή τροποποίηση, η προσαρμογή να γίνει. Οι ε, είναι και επαγγελματίες παίκτες του χόκεϊ και τα λοιπά. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι σημαντικό αυτό πτυχή και το θέμα της ε, ευρωπαϊκής ε, σημαίας καλή ιδέα είναι διότι ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ευχαριστώ. Mr. Σε ευχαριστούμε Μπάγκο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω ουγγρικά. Θα ήθελα να παρέμβω στα αγγλικά, αλλά δεν θέλω να δημιουργηθούν κάποιες παρανοήσεις και για τον συνάδελφο από το Ηνωμένο Βασίλειο στο σημείο 5 για τους χούλιγκαν. Χαίρομαι πρέπει να πω για το ότι αυτό το σημείο σε σχέση με το πρόγραμμα έχει ληφθεί υπόψη, έχει συμπεριληφθεί ο συνάδελφος Σαντιάγο το έχει λάβει υπόψη και το έχει καλύψει. Υπάρχουν αθλήματα που έχουν σημειώσει πρόοδο και σημαντικά μέτρα έχουν ληφθεί. Χαίρομαι γι' αυτό. Μου αρέσει αυτή η έκθεση και εμένα. Πολλοί γνωρίζουν ότι εγώ σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή είμαι μέλος ε, πρόσφατα βέβαια, εδώ και μικρό χρονικό διάστημα. Όμως βλέπω πόση δουλειά έχει επενδυθεί από τον συνάδελφο σε αυτή την έκθεση και πόσο έχουν επενδύσει δουλεύοντα και οι άλλοι συνάδελφοι. Μία σύντομη ερώτηση θα είχα στο σημείο 25 αφορά <clears throat> το θέμα από πλευράς Μπόσκο, δηλαδή να προαχθεί η κινητικότητα. Εδώ ήδη ε, έχει υπάρξει διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Έρασμος για τους αθλητές, για αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα να ρωτήσω, έχει κάποιες απόψεις ο εισηγητής, θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό. Ευχαριστώ. Merci, Madame la Présidente. Je vous... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να θίξω κάτι. Κάτι που δεν έχει απασχολήσει ακόμα αρκετά την Επιτροπή μα, ενώ αποτελεί αρμοδιότητά μας. η εκπαίδευση. Είμαστε και Επιτροπή της εκπαίδευσης και της Παιδείας. Λοιπόν, η παιδεία και η εκπαίδευση στην, ε, στον αθλητισμό για, τις κοινωνικές της, ε, για τα κοινωνικά της ωφέλη θα πρέπει να αποτελεί μέρος ε, του, στο, του εκπαιδευτικού συστήματος των κρατών μελών. Να επανέλθω λοιπόν στην πρόταση ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να είναι δικαιούχος των διευθυντικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως και προωθεί τους ίδιους στόχους με τα διευθυντικά ταμεία, την πολιτική συνοχής ο αθλητισμός. Χρειάζονται λοιπόν και δράσει εκπαιδευτικέ για να προωθηθεί η Ευρωπαϊκή και στον τομέα του αθλητισμού. Και βεβαίω για την Ευρωπαϊκή ημέρα του αθλητισμού, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα για να περάσουν τα μηνύματα τα οποία θέλουμε να μεταδώσουμε. Κάθε χρόνο το να ορίζεται μια Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του αθλητισμού, αθλητισμού μου φαίνεται πολύ καλή ω ιδέα. Και τώρα φαντάζομαι ότι ο Σαντιάγκο δεν ε, προτείνει να δημιουργηθεί αναγκαστικά και να συμμετέχουμε στη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Διατητικού Δικαστηρίου. Ε, είναι μια ιδέα και κάτι που πρέπει να προωθηθεί και για την Ευρωπαϊκή Σημαία νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να προβάλλουμε τις αξίες μας. Ο κ. Σκουρία. Ευχαριστώ. Να πω απλώς ότι η έκθεση αυτή όπως Μα είπε και στι προηγούμενε μα συζητήσει στην Επιτροπή ο Σαντιάγκο, είναι ιδιαίτερα πλήρη. και πολύ καλά συνταγμένη. Να τονίσω εδώ τη σημασία της διάστασης της συμμετοχή των γυναικών. Διότι σκεπτόμενοι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012, να θυμόμαστε ότι σε κάποιε χώρες του κόσμου δεν είναι δυνατόν να αθλούνται οι γυναίκες ελεύθερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν καλό είναι να το υπογραμμίζουμε αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η αξία ισότητας και ελευθερίας. Επίσης, καλό είναι να επισημάνουμε και τη δυνατότητα που έχουν τα διαρθωτικά ταμεία να χρηματοδοτήσουν τη δυνατότητα της άθλησης, την πρόθεση του αθλητισμού μεταξύ εγκαταστάσεων αθλητικών και δεν θα επεκταθώ σε κάτι άλλο πέραν του αθλητισμού Απλώς να πω ότι η Ευρωπαϊκή Σημαία βρίσκεται μπροστά από τα βασικά μέγαρα, τα διοικητικά των εθνικών μας κρατών, τα προεδρικά μέγαρα, τα κοινοβούλια. Δεν βλέπω πρόβλημα να, υπάρχει, να κυματίζει στα γήπεδα. Επειδή έχει περάσει η ώρα, δεν θα μιλήσω. Καλή έκθεση, καλή βάση, θα κάνουμε τροπολογίες και θα συνεχίσουμε. Θαυμάσια. Η κυρία Χάνιβο. Όχι για τη σημαία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω από τη Βρετανική Σκοπιά ότι δεν συμφωνώ με ε, όλους αυτά που λένε. Έχετε δίκιο, Πρόεδρε. Είναι σχέτη πρόταση. Μπορείτε να την απαλείψετε, να κάνετε ένα ε, κείμενο, μια τροπολογία για να διαγραφεί. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το να ε, προωθεί οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ταυτότητα. Θέλω να γραφτεί ε, στα πρακτικά σε αντίθεση με άλλους Βρετανούς βουλευτές και κινδυνεύουμε να χάσουμε ε, πολλά καλά από τα όσα προτείνει η έκθεση. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τον εισηγητή. Είναι εξαιρετική η έκθεση του. Το είπε και ο Μάρκος Κουρία προηγουμένως για τις γυναίκες στον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ δουλειά που μπορούμε να κάνουμε εκεί και να συμφωνήσουμε για αυτό το θέμα ε, για να συνεχίσουμε με επικοδομητική ε, στάση. Και υπάρχει μια τεράστια κοινωνική διάσταση. Δεν μιλήσαμε πολύ για την υγεία ε, και αυτό θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και ο Ούγγρος συνάδελφος είπε κάτι για τη βία και τις διακρίσεις και φοβούμαι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο ποδόσφαιρο έχουμε πολύ κακές επιδόσεις και ε, πρέπει να κάνουμε κάτι διεθνώς και στην Ευρώπη. Και τέλος, του χρόνου θα γίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο Ολυμπιακοί Αγώνες και τέλη Αυγούστου θα τους επισκεφθούμε κιόλας και ελπίζω η επίσκεψή μας να εγγραφεί σε αυτό το πλαίσιο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε τον αθλητισμό και να ξεφορτωθούμε σε αυτές τις γελίες ιδέες που έχουν κάποια μέλη εδώ ότι θέλει να βάλει χέρι η Ευρώπη ε, κάπου στον αθλητισμό να είναι πανευρωπαϊκός ενιαίος. Καμία σχέση. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Πάρα πολύ καλή η έκθεση και την υποστηρίζω ολόψυχα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόκεγκαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επειδή είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό, θα μιλήσω δανεικά. Όπως και ο Πολωνός συνάδελφος έκανε την παρέμβασή του στα πολωνικά. Έτσι και εγώ θα μιλήσω στα σουηδικά στα δανέζικα με συγχωρείτε ευχαριστώ έχει αναφερθεί σε σχέση με την ειδική του ομάδα ο Ισήτη και θέλω να πω σε σχέση με την ειδική μου ομάδα υποστηρίζω την έκθεσή του είναι καλή, είναι σοβαρή καλύπτει όλα αυτά τα οποία είναι αναγκαία μέσα σε αυτό το πλαίσιο και όταν γίνεται λόγο για το άρθρο 165 τη συνθήκη Λισαβόνα, τότε έχουμε μια καλή βάση να δράσουμε με βάση αυτό. Εξ ονόματος της ομάδας μου της Άλντε θα ήθελα να πω ότι εδώ υπό το δικό μου πρίσμα στα ουσιοθέστερα θέματα πρόκειται για την κοινωνική, κοινωνική διάσταση του αθλητισμού να υπάρξει συνοχή και συνεκτικότητα που θα δημιουργείται, να έρθουν σε επαφή οι πολίτες, η δημόσια υγεία να είναι ένα κέριο κεντρικό σημείο σε αυτό το πλαίσιο και πιστεύω ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την συνεκτικότητα και συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα δημόσιας υγείας εκεί πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα τον αθλητισμό τον θέσουμε στο προσκήνιο στην πρώτη γραμμή και να τύχει ιδιαίτερης προσοχής Πρέπει με την κυρία Μακλάκη εδώ να πω ότι συμφωνώ έχει δίκιο σε αυτό το σημείο παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι πρέπει να προσέξουμε αυτά τα πολύ συναισθηματικά φορτισμένα θέματα να μην ξεκινήσουν μια ευρύτερη αντιπαράθεση για ύμνους, ε, ε, σημαίες και τα λοιπά. Πολύ συχνά οι πολίτες έτσι αποκτούν μια αποθούνται και υπάρχει και λαϊκισμός, λαϊκίστικη τάση που εκμεταλλεύονται κάποιοι. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα δύσκολο πεδίο όταν συζητάμε για τέτοια θέματα όπως για σημαίες. Στην Δανία υπήρξε ένα παρόμοιο άρθρο. Πρόκειται πραγματικά ουσιαστικά για το ίδιο άρθρο όπως εκείνο στον Βρετανικό τύπο. Και είναι μια σφιγμομέτρηση, ένα ερωτηματολόγιο που δείχνει ότι οι πολίτες πιστεύουν κατά 80% ότι είναι μια, ε, κάτι το παράλογο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το λάβουμε υπόψη ε, αυτό το πράγμα και συμφωνώ από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι φυσικά μια τέτοια πρόταση μπορεί κανείς να την καταθέσει. Εθελοντικό θα είναι το πλαίσιο της εφαρμογής. Μπορεί και να το διαγράψει κανείς, να το απαλείψει αν δεν επιθυμεί να το ακολουθήσει. Αλλά όταν πρόκειται για τον αθλητισμό, για θέματα αθλητισμού πρέπει τέτοια πράγματα να λαμβάνονται υπόψη, να μην αφήνουμε ευκαιρία στους λαϊκιστές στον λαϊκισμό να παρισφραίει και να παραλύει τα πράγματα και να τα υπονομεύει. Γιατί αν παραμείνουν αυτά τα πράγματα έτσι, τότε αυτό θα είναι το κυριότερο σημείο αντιπαράθεση και δεν υπάρχει κανένα λόγο να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στου λαϊκίστες. Κατά τα άλλα συμφωνώ με την έκθεση. Σκέλη, παρακαλώ. Είναι πολύ σύντομα. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που είπατε κι εσείς και η κυρία Χάνιμπολ για το βρετανικό τύπο να το έχει υπόψη του. Είναι πρόταση, είναι μια σύσταση. Αυτή είναι η δουλειά του εισηγητή, να κάνει προτάσεις, εμείς συζητούμε και αποφασίζουμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι το 50% των Βρετανών θέλουν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας εκπλήσει με όλη αυτή την αρνητική προβολή και την παραπληροφόρηση για τα όσα συμβαίνουν. Και εμείς δεν τονίζουμε αρκετά τα καλά μας. Είμαστε οι χειρότεροι διαφημιστές ε, και εκπρόσωποι δημοσίων σχέσεων. Όταν μας επιτίθενται δεν αντιτιπιθέμεθα και ε, αφήνουμε να δρουν έτσι διάφορα στοιχεία του βρετανικού τύπου. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Τζον. Όλοι γνωρίζουν ότι στη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει δυνατότητα να σηκωθεί κανείς να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι απλώς για να το ξέρουμε. Λοιπόν, ήθελα να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, στα γερμανικά. Στην έκθεση αυτή θα ήθελα να προσθέσουμε το εξή ακόμα. Ότι θα πρέπει να σκεφτούμε το εξή γεγονός. Να μην υφίσταται διακρίσει οι γυναίκε στο ποδόσφαιρο. Με την εξή έννοια, την πολύ συγκεκριμένη. Οι Ολυμπιακοί κανόνες ορίζουν τι φοράει κανείς, έτσι, αθλητής. Είναι οι Ολυμπιακοί κανόνες αυτοί. Όλοι το ίδιο. Σόρτ, φανέλα, τα γράφουν ε, ρητά. Ε, σε κάθε ε, άθλημα υπάρχει αντίστοιχη αμφίεση. Και στο μεταξύ τι κάνουν χώρες όπως το Ιράν. Εφήβραν ότι θα πρέπει κανείς να είναι τυλιγμένος εντελώς, η γυναίκα δηλαδή, και τότε επιτρέπονται. Εντάξει, να επιτρέπεται, αλλά αυτό που οδηγεί ότι στις χώρες αυτές τις Ισλαμικές, οι γυναίκες που τόλμησαν μέχρι τώρα να κάνουν κολύβεις ας πούμε με το κανονικό μαγιό ή να αγωνίζονται με την κανονική φανέλα χωρίς να είναι τυλιγμένες στα φασκές δεν ε, τολμούν να το κάνουν γιατί δεν τις αφήνουν να συμμετέχουν πρέπει να είναι καλυμμένες από πάνω μέχρι κάτω. Και ντράπηκα, ε, η γερμανική εθνική ομάδα γυναικών έχασε βέβαια, αλλά πήγε στο Ιράν και έπαιξε σε μια τέτοια ποδοσφαιρική διοργάνωση. Στο Ιράν έγινε με άλλες ομάδες από Ισλαμικές ε, χώρες σε ένα τέτοιο ποδόσφαιρο ε, και πρωτάθλημα και βάλαν και οι Γερμανίδες φερετζέ για να παίξουν ποδόσφαιρο. Έτσι λέω, μα πάτε καλά σας έχει στρίψει καμιά βίδα, τίποτα. Ε, θα πρέπει να το πούμε παντού. Υπάρχει αμφίεση συγκεκριμένη επίσημη από του Ολυμπιακού Αγώνε. Δεν χρειάζεται να πούμε για μουσουλμάνες ή μη, ό,τι λένε οι Ολυμπιακοί κανόνε. Και να γράψουμε και στη FIFA και σε όλου αυτού που ενέχονται να φροντίσουν οι γυναίκε που τολμούν να βγουν από τον κέτο και δεν καλύπτουν το κεφάλι και το πρόσωπό τους, να μην τους αναγκάζουν να δεχόμαστε ε, να είναι καλυμμένες από την κορφή ως τα νύχια για να παίξουν ποδόσφαιρο. Τα λέω γιατί εξοργίστηκα τόσο πολύ που ήθελα να τα βγάλω από πάνω μου. Δεν ξέρω, μήπως έχεις και εσύ καμία ιδέα πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Α, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να πει τίποτα σχετικά. Ποιο θέλει το λόγο από την Επιτροπή. Εγώ. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον εισηγητή για πραγματικά μια περιεκτική πλήρη έκθεση και εκτιμούμε ιδιαίτερα και τις προτάσεις που ε, μπορούν να αποτελέσουν ε, θέματα προβληματισμού. Ευχαριστούμε διότι αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και την οτροπία και τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό όπως ε, προβλέπετε και αντανακλάτε στη συνθήκη αυτό το θέμα υπογραμμίζει η έκθεση τις σημαντικές αξίες και αρχές ε, που είναι εγγενείς στον αθλητισμό, τονίζει τις ε, μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και υπογραμμίζει και αυτό είναι κέρια σημασία και εδώ διαφωνώ κάπως ε, μαζί σας υπογραμμίζει και λέει ότι ο αθλητισμός συνεισφέρει αυθεντικά στο πλαίσιο της στρατηγικής για τους στόχους για την Ευρώπη του 2020 και τη στρατηγική αυτή. Είναι ισορροπημένη η έκθεση. Καλύπτει τις διαφορετικές πτυχές και παραμέτρους του αθλητισμού, την κοινωνική, την οικονομική και την διοργανωτική πτυχή για τα θέματα του αθλητισμού και εξετάζει τον τομέα σύνολο και για τον επαγγελματικό και τον εραστεχνικό αθλητισμό. Έτσι λοιπόν συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει τις γενικές κατευθύνσεις αυτής της έκθεσης που σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμίζονται με την ανακοίνωσή μας από πλευράς μας. Έχουμε διαφορετικές προτάσεις στην έκθεση και μπορούν κάποιες από αυτές να εξεταστούν ή να συνδεθούν με τις δράσεις που αναπτύσσονται από πλευράς του ψηφίσματος του Συμβουλίου για τον Αθλητισμό της 20ης Μαΐου που εγκρίθηκε στις 20 Μαΐου και μπορούν τώρα στις νέες ε, οργανωτικές και εργασιακές δομές να ενταχθούν και να προχωρήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει λοιπόν σε αυτό το έργο και θα βοηθήσει στην εφαρμογή και υλοποίηση κάποιων προτάσεων και σίγουρα εκείνων των προτάσεων που εμείς διατυπώσαμε στην ανακοίνωσή μας. Μεταξύ άλλων θα δημιουργήσουμε κάποιες μελέτες που θα συνταχθούν σύντομα αναφέρομαι στα παιδεία στους τομείς είτε είναι πολύ πρόσφατες μελέτες που ξεκίνησαν από εμάς είτε θα ξεκινήσουν σύντομα και βρίσκονται υπό προετοιμασία μια μελέτη που μόλις ξεκίνησε για την εθνική νομοθεσία όσον αφορά την απάτη της ε, απάτης στον αθλητισμό σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή στημένα παιχνίδια και εκδηλώσεις. Υπάρχει η ιδέα επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα του να προταθεί μια σύσταση από πλευράς του Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου για την δημιουργικότητα και αυτή η μελέτη θα ξεκινήσει, θα συνταχθεί πολύ σύντομα. Επίσης μια μελέτη, μια μελέτη για τις μεταφορές παικτών, εξαγορές και μεταφορές από τη μία στην άλλη ε, ομάδα παικτών. Θα ξεκινήσουμε και μια μελέτη για την εποπτεία των ε, αθλητικών εκδηλώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια και μετά μια μελέτη για το τι θα μπορέσει να γίνει για την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσα στο πλαίσιο του αθλητισμού στην ΕΕ. Σύντομα τώρα στη συνέχεια δύο παρατηρήσεις. Τίνο βλέπετε κάπως να διαφωνήσω κάπως με την κατεύθυνση της έκθεσης, ιδιαίτερα με τις παρατηρήσεις του εισηγητή για το μέλλον όσο αφορά την υγεία διότι αναφέρεται ότι η υγεία και ιδιαίτερα οι σωματικές δραστηριότητες ε, δεν είναι ή δεν θα έπρεπε να είναι μείζον θέμα για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ διαφωνούμε κάπως σε σχέση με την ανακοίνωσή μας όπως προαναφέρεται. Εμείς ε, σε σχέση με τις δράσεις που προτείνουμε και με τις προκαταρκτικές δράσεις που χρηματοδοτούμε στον τομέα του αθλητισμού π.χ. για το 2009 στον τομέα του, της υγείας είναι σημαντικό να υπάρξει έργο που θα αναλάβουμε ε, πέρα από τα εθνικά σύνορα. Και ένα άλλο σημείο επιπλέον θέματα για τα διαθροτικά κονδύλια των διαθροτικών ταμείων. Ε, εργαστήκαμε σκληρά με τους συναδέλφους στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε ο αθλητισμός να διασφαλιστεί ότι θα ενταχθεί και στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο και πράγμα το οποίο τώρα συζητείται στους κανονισμούς για τα ταμεία και τη διάθεση των κονδυλίων τους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και δύο λόγια τελευταία, όπως προανέφερα, για την πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω του αθλητισμού και των αθλητικών δραστηριοτήτων. Όπως γνωρίζετε γενικά, ναι μπορούμε να πούμε ταυτότητα και ευδιάκριτος χαρακτήρας για τη σημαία είναι κάτι σίγουρα που δεν είμαστε εναντίον αυτού. Αλλά και πάλι με επίμαχο αμφίσιμο τρόπο συζητείται και δεν είναι δεδομένη η έκβαση στα όργανα και προσβλέπουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση. Ευχαριστώ Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχετε διαβάσει την έκθεση στο πλήρες εύρος όταν λέτε ότι είπε ο εισηγητής ότι τα αθλήματα δεν διαδραματίζουν ρόλο για την υγεία. Εγώ τη διάβασα. Ίσως ο ίδιο ο Σαντιάγο μπορεί να πει κάτι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε για Ο κύριος Φίσα και πάλι στο τέλος για να ολοκληρώσουμε. Αυτό το θέμα θα το αφήσουμε στο περιθώριο όμω, εντάξει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Στο τέλος θα πω κάτι για τη σημαία, αλλά ε, αρχικά το εξής και το λέω για τους συναδέλφους κυρίως που είναι καινούργοι και ήρθαν πρώτη φορά στην Επιτροπή μας. Επανειλημμένα έχω επαναλάβει ότι η έκθεση αυτή και ο αθλητισμός γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο σύνορα πολύ ξεκάθαρα. Την αρχή της επικουρικότητα και την αρχή της ιδιαίτερότητα του κάθε αθλήματος. Το έχω ξαναπεί επανειλημμένα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Πρώτον, εγώ έχω διατελέσει στην Ισπανία ε, υφυπουργός αθλητισμού και οι αρμοδιότητε δεν είναι μόνο τη κεντρική κυβέρνηση πλέον, αλλά είναι αρμοδιότητε των αυτονόμων περιφερειών πλέον. Και ξέρω πολύ καλά ότι οι δικές μου αρμοδιότητε, και ακόμα και σε κρατικό επίπεδο, ήταν πάρα πολύ περιορισμένες. Λοιπόν, α μην μιλήσουμε τώρα καν για τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητε. Κάτι άλλο που είπε πολύ ωραία η κυρία Πακ είναι ότι από πολλές ενώσεις, ομοσπονδίες, συλλόγου ευρωπαϊκούς έρχονται και μας ζητούν να ρυθμίσουμε κάτι στην Ευρώπη γιατί υπάρχει ανάγκη. Αυτό μας το ζητούν οι ίδιοι και αυτό φρόντισα να κάνω. Η ιδιαιτερότητα από την άλλη. Εγώ προέρχομαι από τον αθλητισμό. Είναι πολύ βρετανικό το σπόρ μου, ε, ε, πολύ κλασικό, είναι το γκολφ. Ήμουν στην εθνική ομάδα της Ισπανίας του γκολφ Είμαι και μέλος ε, της Βασιλικής Λέσχης Γκολφ του Σεντ Άντριους. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι ιδιαιτερότητα έχει το κάθε άθλημα και ο αθλητισμός και πώς ε, σκέπτονται οι Βρετανοί για τον αθλητισμό. Αλλά επίσης να πω και το εξής είναι ιδιαίτερο το σπορ, αλλά και ο αθλητισμό όπως κανένα στον κόσμο δεν είναι υπεράνω του νόμου. Και θα πρέπει να το τονίσουμε και πάλι. Εντάξει, είναι κάτι ιδιαίτερο ο αθλητισμός, αλλά θα πρέπει αναπερίπτωση να το μελετούμε και δεν είναι γενικός κανόνας, δεν είναι καμία βούλα του Πάπα α πούμε, που έχει το αλάθητο και κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Ε, πολλές ιδιαιτερότητες υπάρχουν και σε αυτό το θέμα. Δύο πράγματα ακόμα. Ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός στη διατύπωσή μου. Και για τη σημαία την ευρωπαϊκή ας πούμε, ε, μιλώ για τη σημαία αυτή επιπλέον των ε, διαφόρων ε, εθνών, κρατών και εννοώ και τη φανέλα και στη Βρετανία προτείνει, προτείνει λέει, προτείνει, δεν είναι υποχρέωση. Όποιος δεν θέλει μην το κάνει και δεν τρέχει τίποτα και πάλι ωραία είμαστε. Εγώ είμαι ακρεφνής ευρωπαϊστής. Δεν ξέρω για τους άλλους. Δική μου έκθεση είναι επιτρέψτε μου να το προτείνω, με τι άλλο. Και κάτι ακόμα, κυρία Μακλάρκιν, υπάρχει μια αντίφαση όταν λέτε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό στη βάση του. Μα ε, τότε μπαίνουμε εκεί στα χωράφια και τις αρμοδιότητες των κρατών και των περιφερειών, αν φτάσουμε στη βάση του αθλητισμού. Είναι πολύ καλό να προωθείται ο αθλητισμό, αλλά αυτό είναι δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης των περιφερειών και των κρατών. Δεν είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιότητα. Να υποστηρίζουμε, να προωθούμε, αλλά αυτό θα παραπήγαινε πραγματικά και θα ήταν κατά τη αρχή τη επικουρικότητας. Γιατί ανταγωνίζεται ακριβώ τι αρμοδιότητες των οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση ο αθλητισμό στη βάση. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να τον υποστηρίξουμε, αλλά το πώ πρέπει να το αποφασίζουν οι ΟΤΑ. Οπότε βλέπω μια αντίφαση σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σα ευχαριστώ όλου για τα σχόλιά σα. Αν μου επιτρέπετε ένα που ακούστηκε επανειλημμένα και η κυρία Μποσκούρτ το είπε και άλλη, ε, για το διαιτητικό δικαστήριο. Το είπε πολύ ωραίο ο κύριος Μπελέτ. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ το εξής. Όταν κάποιος έχει ένα θέμα με το ντόπινγκ, ας πούμε, του επιβάλλεται μια κύρωση αθλητική. Από μια ομοσπονδία κανονικά. Και ο αθλητής αυτός δεν είναι αθλητές, είναι ε, αγωνιζόμενοι, δεν ξέρω πώς να το πούμε πάντα, είναι παίκτες. Εν πάση αυτός ο αθλήτης ε, τελικά πηγαίνει στο ανώτατο δικαστήριο ε, το διαιτητικό, το αθλητικό στη Λοζάνη. Αν διαφωνεί με την άποψη αυτή, όπως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ε, προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη, σε ένα αστικό δικαστήριο. Και μπορεί να υπάρξει κάποια περίπτωση όπου να διαφέρουν οι αποφάσεις. Υπήρξε και η υπόθεση με τα Μετίνα που είχε καταδικαστεί ε, ε, σε δύο χρόνια ε, αποχής από τον αθλητισμό. Το επόμενο δικαστήριο, το πολιτικό, τον δικαίωσε. Αλλά στο μεταξύ είχε χάσει το τρένο γιατί είναι πολύ σύντομη η σταδιοδρομία επαγγελματική ή άλλη ενός αθλητού. Λοιπόν, να υπάρχει κάτι στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει στο το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο που είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο της ε, Ελβετίας. Επίσης υπάρχουν άλλα παραδείγματα, Αυστραλία, Ηνωμένε Πολιτείε, ισχύουν αυτά. Ε, έγινε λόγος για τα διαρθρωτικά ταμεία, για τις γυναίκες, πολύ σημαντικό αυτό, από κάθε άποψη. Το έχω εντοπίσει το πρόβλημα κι εγώ. Η λύση δεν είναι εύκολη Ούτε είμαι σύμφωνος με ποσοστώσεις και υποχρεωτικό αριθμό γυναικών στις αντιπροσωπείες, στους συλλόγους, στις ε, ομοσπονδίες. Και βεβαίως ε, σημειώνω αυτό που είπε η κυρία Πακ. Να βρούμε ε, ένα τρόπο με τροπολογία, συμφωνώ, για να αποφύγουμε αυτό το είδος καταναγκασμού των γυναικών ε, να φοράνε φούστες, ισλαμικά μαντήλια, δεν ξέρω, όχι μόνο στους ολυμπιακού Αγώνες, παντού. Και είναι και κατά του πνεύματο του αθλητισμού. Δεν καταλαβαίνω αυτό που είπε για την Υγεία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην αιτιολογική σκέψη Β λέει λαμβάνοντα υπόψη ότι ο αθλητισμό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υγεία στη σύγχρονη κοινωνία και ένα βασικό συστατικό τη ποιοτική εκπαίδευση. Το λέει η αιτιολογική σκέψη Β. Και λυπάμαι που δεν μπόρεσα για λόγους χρονικούς να μην εξηγήσω όλα αυτά που ήθελα. Όποιος αθλείται κάνει τεράστιες οικονομίες ε, στις ε, δαπάνες υγείας ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα λοιπόν. Μπορούμε να τα συζητήσουμε. Τα βασικότερα όμως είναι σαφή νομίζω. Ευχαριστώ η Πρόεδρος. Γεγονός είναι ότι στην αιτιολογική σκέψη Β αναφέρεται η υγεία και διαβάστε και την αιτιολόγηση του συναδέλφου. Στην αιτιολογική έκθεση έχει ολόκληρη παράγραφο. Ένα πρόβλημα έχει μόνο ο αγαπητό συνάδελφο είναι ότι μπορεί να είναι σύντομη η έκθεσή του. Εμεί μπορούμε να την κάνουμε πιο μακροσκελή με επιπλέον τροπολογία για την υγεία. Να σκεφτούμε και αυτό. Μα το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία. Τώρα, Είπαμε ότι δεν θέλουμε η προθεσμία να είναι στις 31 Αυγούστου, αλλά 6 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, αλλάζει η προθεσμία για τις τροπολογίες, αντί για τις 31 Αυγούστου, 6 Ενάτου. Ωραία, σας ευχαριστώ. Καταπληκτική συζήτηση. Πάντα εμπλουτίζεται από έναν που είναι μονίμως από αλλά και από άλλους. Πάμε στο 14 τώρα, που δεν θα σας ενδιαφέρει τόσο πολύ γιατί λέει η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, όλα τα τμήματα. Κύριε Λόκεγκαρτ, έχετε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος, Πρόεδρε. Οι προτάσεις της εκθεσής μου έχουν εξεταστεί και ήδη ψηφίσαμε και προ λίγο, όπως θα βλέπετε λοιπόν όλοι. Υπάρχουν α, τέσσερα σημεία. Ένα για τα εκπαιδευτικά συστήματα, έπειτα για τη διαβίου μάθηση, μετά για τον αθλητισμό. Το θέμα μετά του αποθεματικού και μετά τα ευρωπαϊκά σχολεία. Όλα αυτά έχουν καλυφθεί. Υπήρξαν σχετικές προτάσεις. Και οι, μου, οι δικές μου προτάσεις έχουν καλυφθεί σε τρεις τουλάχιστον από αυτούς τους τίτλους στη συζήτηση περί υπερπολογισμού. Άλλη, μα. You want, please. Θέλετε εσείς να παρέμβετε παρακαλώ. <laughs> Um, I've made my comments before. Έκανα και προηγουμένως τα σχόλιά μου. Απλώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν δεπανούμε τα χρήματα άλλων. Είμαι ικανοποιημένη πάντω με όσα έκανε ο κύριο Λάκεγκαρτ. Έχει ανοίξει τη συζήτηση ακόμα και στο να συμπεριλάβει τα δικά μου, ή να ακούσει τουλάχιστον τα δικά μου σχόλια. Για τον αθλητισμό, λέγαμε για 8 εκατομμύρια για τον αθλητισμό. Εγώ ήθελα στον προπολογισμό να εξοικονομήσουμε με τι δικές μου προτάσεις 152 και να ευθυγραμμίσουμε λίγο τι προτάσει μα για, το πόσο χρήματα, για το πόσα κονδύλια ζητούμε. Γιατί έχω δίνουμε πάντα την εντύπωση ότι εύκολα θα πάρουμε τα χρήματα άλλων. Ναι, αλλά μια στιγμή πρόκειται για τα παιδιά μα, έτσι. Για τα παιδιά μα πρόκειται. <clears throat> Αν έχετε εσεί παιδιά και για τα δικά σα τα παιδιά, για το μέλλον του πρόκειται. Ένα πολύ μικρό τμήμα του προπολογισμού έχουμε. Εμεί για το λάδι, για το ελαιόλαδο δίνουμε περισσότερο από ό,τι για την παιδεία και την εκπαίδευση. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσει, αλλά να κάνουμε αλλού, όχι στην εκπαίδευση και παιδεία και κατάρτιση. Σε αυτά τα θέματα πρέπει περισσότερα να δίνουμε. κυρία Παλιαδέλη παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, έχουμε ήδη συνεργαστεί με τον κύριο Λόκεγκαρτ πολύ καλά στη φάση της, των παρατηρήσεων για τον προπολογισμό και τις προτάσεις μας. Η μία μόνο παρατήρηση την οποία την έχω κάνει και προσωπικά. Πιστεύω ότι στο σύντομο κείμενό του λείπει ένα πολύ βασικό κομμάτι, σχόλιο που αφορά στον πολιτισμό, αλλά θα μας δοθεί φαντάζομαι η δυνατότητα με τις τροπολογίες μας να συμπληρώσουμε αυτό το κενό. Ενώ μιλάμε για παιδεία για αθλητισμό πολύ για δημοσιογραφία και μέσα ενημέρωση. λείπει εντελώ ο πολιτισμό. ελπίζω με τροπολογίε μας να καλύψουμε αυτό το κενό γιατί θεωρώ σημαντικό να αναφέρεται ως, όταν αναφέρεται ως εργαλείο για τη συνοχή να χρηματοδοτείται, να και αναλόγως. Ευχαριστώ. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, μόλις είπατε ότι υπάρχουν πολλοί τομείς όπου είστε υπέρ των οικονομιών. Θα μπορούσατε λίγο να το διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε. Ε, όχι τώρα. Γιατί ε. τώρα συζητάμε για το δικό μας προϋπολογισμό και θέλω να αυξηθούν τα κονδύλια. Σε άλλη επιτροπή θα πάρω θέση. Μα πήρατε μαζικά θέση. Όχι, εξήγησα ότι δεν θέλω τους τομείς που αφορούν την επόμενη γενιά, την παιδεία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό. Δεν θα κάνουμε περικοπές εκεί, να αυξήσουμε τα κονδύλια. Και εδώ σταματώ. Ε. Και δεν χρειάζεται να σας δώσω λογαριασμό ε, για το πού θα περικόψουμε. Υπάρχουν πολλά, αλλά δεν είναι της παρούσης επιτροπής. Ο συνάδελφος Μπελέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Συμφωνούμε με το σχέδιο έκθεση όπω το έχει συντάξει ο εισηγητή. Απλώ μια παρατήρηση για το σημείο 3. Η διατύπωση είναι κάπω επικριτική και αρνητική μάλιστα. σω να το αναδιατυπώναμε για να πούμε το ίδιο, μεταδιατυπώνοντα το με τρόπο πιο θετικό. Να ζητήσουμε από την Επιτροπή να καταβάλει περισσότερε προσπάθειε για τα μέσα μαζικής επικοινωνία στην επικοινωνία και αυτό να γίνει σαφές προ όλου. Ε, ε, Σε ό,τι αφορά τα δύο πρώτα σημεία για τη δική μας γενική διεύθυνση, τη διαβίωμάθηση και τον αθλητισμό, για το κατά πόσο μπορεί να προβλεφθεί, θα προβλεφθεί μάλλον διπλασιασμός του κονδυλίου ε, του σχετικού για το διάστημα των ερχόμενων πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών. Και τέλος πάντων, αν συγκρίνουμε τις επταετής περιόδους, η αύξηση που προτείνεται είναι 70%. Και μάλιστα θα δοθεί και μεγαλύτερη προβολή στον ερχόμενη περίοδο προγραμματισμού. Μέχρι το 2020 μάλιστα προβλέπεται να υπάρξει υπερδιπλασιασμό σε σχέση με το 2013. Με τις προτάσεις λοιπόν της Επιτροπής θα δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση να την περαιώσουμε εδώ, να την ολοκληρώσουμε. Στις 6 Σεπτεμβρίου έχουμε και για αυτό το θέμα εκπνοή προθεσμίας για τις τροπολογίες. Κύριε Λόκεγκαρτ, θέλετε να πείτε κάτι. Κύριε Λόκεγκαρτ, όχι, εντάξει, ωραία. Περνάμε στο σημείο 15. Αλλά κύριος Μιγκάτσκι δεν είναι πια παρόν στην αίθουσα. Ναι, είναι. Εντάξει, ωραία. Εκρίμα τότε. Λοιπόν, μια νέα απάντηση για την πολιτική γειτονία ε, που αλλάζει. Ευχαριστώ. Ε, Δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο σύντομη η εξέταση της προηγούμενης έκθεσης. <laughs> Κάτι που το συζητήσαμε και με την κυρία Νευντάλοβα. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι πολύ σύντομη. Υπάρχει λίγος χρόνος στη διαθεσή μας. Παρακαλώ όλοι να το έχετε κατά νου. Θα πρέπει γρήγορα να διοριστούν οι σκιώδεις συζητητές για να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Υπάρχουν και κάποιοι αντικειμενικοί περιορισμοί. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο η έκθεσή μου επικεντρώνεται σε έξι μόνον σημεία. Θα τα παρουσιάσω συνοπτικά. Στο πρώτο σημείο ζητάτε κατανομή, ισότιμη κατανομή των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Εδώ έχουμε κατά νου την Βόρεια Αφρική. Στην τελευταία περίοδο κρίσης, κατά τη λεγόμενη δηλαδή Αραβική Άνοιξη και τις επαναστάσεις της ε, χώρες της Βορείου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίθηκε στο ύψος των περιστάσεων οι πολίτες που κατοικούν σε χώρες με καθεστώτα μη δημοκρατικά προσδοκούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει για να προασπιστεί τις κοινέ μας αξίες. Η αρχή αυτή λοιπόν, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να εφαρμόζεται και στους ε, γείτονε ή εταίρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ Ανατολά ή προ τον Νότο. Έχουμε και εκεί χώρε μη δημοκρατικέ, όπω η Λευκορωσία, α πούμε. Θα πρέπει και οι πολίτε των χωρών αυτών να μπορούν να επωφεληθούν από την στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο σημείο. Ζητούμε απλουστεύσεις, απλουστεύσεις για τις σπουδέ και τους νέους φοιτητέ σε χώρε που τι καλύπτει, τις καλύπτει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία. Πρόκειται για χώρε με τι οποίε συνεργαζόμαστε και του νέου των χωρών αυτών θέλουμε να του στηρίξουμε, στηρίζοντα την ε, κινητικότητα, τι ανταλλαγέ, τι φοιτητικέ, την... τα ταξίδια των νέων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η τεχνογνωσία μας να είναι διαθέσιμη και στους νέους των χωρών αυτών, των ε, χωρών που καλύπτει η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Επίσης, στο σημείο 3 αναφέρεται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας η δημιουργία ενός ε, συστήματος, ενός προγράμματος ανταλλαγών. Κάτι που ήδη προβλέπεται στη Σλοβενία ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Σλοβενική Κυβέρνηση. Όμως, θα πρέπει η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων να είναι όσο το δυνατόν αποδοτικότερη. Με τη δημιουργία ενός ε, πανεπιστημίου, λοιπόν, αυτού του είδους, θα μπορούσαμε να αποσπάσουμε ωφέλη και να ε, γίνουν τα ωφέλη αυτά φανερά και στους, στις χώρες που είναι υποψήφιες για την προσχώρηση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σημείο 4 και 5 ε, επανέρχομαι σε όσα είχα πει στο 2, δεν θα τα επαναλάβω. Στο τελευταίο σημείο ζητούμε στήριξη της ε, κοινωνίας των πολιτών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κυβερνητικών οργανώσεων, ώστε να προαχθούν τα δημοκρατικά συστήματα στις χώρες που βρίσκονται προς Ανατολάς, της Ένωσης και προς τον Νότο. Έδωσε ήδη το παράδειγμα της Λευκορωσίας. Ξέρουμε ότι η διαδικασία προσχώρησης της χώρας αυτής έχει ανασταλεί Έχουμε πολλές απαιτήσει λοιπόν από τους πληθυσμούς αυτούς. Τους ζητάμε να εμπνέονται από τις κοινέ μας αξίες ελεύθερο ελεύθερος τύπος, ελευθεροτυπία δηλαδή, ελεύθερη έκφραση, δημοκρατία. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Εδώ ε, Επίση θα υποβληθούν προφανώ τροπολογίε, υπολογίζω στη συνεργασία όλων σα. Θα τα συζητήσουμε όσα σημεία προκύψουν και δημιουργούν δυσκολίε με του και εισηγητέ. και Ήδη έχουμε σκιώδη εισηγητή από του σοσιαλιστέ. Ελπίζω και οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε να διορίσουν σύντομα του εισηγητέ του, ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε αμέσω μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ για το θέμα αυτό. Οι προθεσμίε πραγματικά είναι φωνικέ.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 είναι πάρα πολύ κοντινέ ε, μετά τα όσα προέβλεψε η Επιτροπή ιστορικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Είμαι ανοιχτό στι παρατηρήσει σα. Ευχαριστώ. επιτρέψτε μου να σα πω κάτι. Ξέρετε ότι δεν είμαι φίλη των γραπτών δηλώσεων και διακηρύξεων. Υπάρχει όμω μια γραπτή δήλωση που μα υποχρεώνει για τι γειτονικέ χώρε την διαβίω εκπαίδευση να την ξεκινήσουμε με προγράμματα. Εγώ δεν θα προσυπογράψω κάτι τέτοιο. Εδώ πρέπει να το κάνουμε. Διότι για αυτό το σημείο το 2 πρέπει να το καταστήσουμε πολύ σαφέστερο. Το 2 θα ήθελα να λέει ότι ζητεί από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι enables και τα λοιπά, αλλά ζητείτε να ανοίξει η διαδικασία της διαβίου εκπαίδευσης και μάθησης προς τις χώρες της γειτονίας, τις γειτονικές χώρες αυτό είναι αυτό που πρέπει να πούμε. Είναι καλύτερο και να μην πούμε μόνο οι φοιτητέ στο Education Europe. Καλύτερο θα ήταν να άνοιγε αυτή η δυνατότητα. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη γραπτή δήλωση. Αυτό σημαίνει έρασμος για, το να πούμε έρασμος για όλα θα ήταν κάτι υπερβολικό. Αυτό όμως εδώ είναι εντάξει, είμαστε ευθυγραμμιζόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Καθήκον μας είναι να προχωρήσουμε έτσι και όχι για μια γραπτή δήλωση που θα πάει στην κάλαθο των αχρήστων. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να δράσουμε ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι. Θα το κάνετε εσείς, αλλιώς θα καταθέσουμε μια τροπολογία αν συμφωνείτε μπορείτε εσείς να το αναλάβετε. Η κυρία Στέρμερα Λόγα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και θέλω να υποστηρίξω τον εισηγητή στο αίτημα αυτό και θέλω και εγώ να πω ότι υπάρχει πολύ λίγος χρόνος και πρέπει να προσέξουμε ή να ανταποκριθούμε σε σχέση με το αίτημα του συναδέλφου. Το ότι βρισκόμαστε υποπίεση χρόνου είναι άδικο όμως. Πρέπει να το επανορθώσουμε. Είναι γνωστός ο εισηγητής ότι ασχολείται με την πολιτική για τη γειτονία και έχει ξεχωριστές θέσεις από πλευράς του και το βλέπουμε και με αυτή την πρόταση. Είναι πολύ σημαντικό, έχει ε, αναφερθεί αρκετές φορές, πρόκειται για την κινητικότητα, μεγαλύτερη κινητικότητα όσον αφορά τις γειτονικές χώρες. Πρέπει να υποστηριχθούν αυτές οι χώρες, όπως κοινά προγράμματα, όπως ο Erasmus Mundus πρέπει να προαχθούν, συνεργασία με πανεπιστήμια πανεπιστήμια, πρόγραμμα Tempus. Πρέπει και είναι θετικό να ανταλλάσσουμε πληροφορίες μέσα σε αυτό το σύστημα μεταξύ των κρατών μελών και μέσα από τα, στα γειτονικά κράτη και κάποια μέρα ίσως αυτά τα κράτη, τα γειτονικά κράτη γίνουν υστερότερα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο διάλογος να γνωρίζουν τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει ε, μια ε, συγκεκριμένη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Πρέπει να, για τη μετανάστευση για παράδειγμα πρέπει να συνεργαστούμε και να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε ισότιμοι και οι διαφορέ δεν θα είναι πολύ μεγάλε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, έχω πολύ λίγο χρόνο. Εμεί ω ομάδα θα καταθέσουμε τροπολογίε, αλλά και με τον εισηγητή θα έρθουμε σε επαφή. Σε επαφή. Του εύχομαι ότι το καλύτερο. Ευχαριστώ. Um, uh, Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί δύσκολο είναι με τόσου λίγου χαρακτήρε να εκφράσει κανεί τόσε ιδέε. Να πω ότι εμεί ενδιαφερόμαστε για τον τομέα τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία στα προγράμματα τη πολιτική γειτονία, διότι είναι ένα τρόπο αυτό να φέρουμε πιο κοντά του πολίτε με μικρές, μικρές εμβέλειας πολιτικές, με συγκεκριμένες δράσεις στην καθημερινή ζωή της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό θα μπορούσε να μας προσφέρει μια προστιθέμενη αξία ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Γιατί Νομίζω ότι αυτά είναι τα πραγματικά μέσα για να αναπτυχθεί η δημοκρατία. Και στον τομέα της διακυβέρνησης και των διοικήσεων, των διοικητικών αρχών. Η πρακτική εξάσκηση μπορεί να ωφελήσει πολύ τις χώρες αυτές και θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το σκέλος να το προωθήσει. Είναι μόνο 10% της πολιτικής γειτονίας. Μάρκο. Ευχαριστούμε κύριο Σκουρία. Ευχαριστώ πρόεδρε κατεύθυνση που έχει δώσει ο συναδελφός και στην έκθεση αυτή είναι πολύ κατάλληλη. Νομίζω ότι και οι αναφορές στην Μεσόγειο, ιδίω για το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο, είναι ένα από τα στοιχεία που ιδιαίτερα θετικά τα βρίσκουμε, διότι αυτό έρχεται να συμπληρώσει και τι δράσει μα στην Ευρωμεσογειακή Συνέλευση. Και για τα προγράμματα κινητικότητας, συμμερίζομαι τις απόψει σα. Οπότε με κάποιες τροπολογίες, κάποιες προσθήκες που πιστεύω πρέπει να γίνουν, θα φροντίσουμε να τις υποβάλουμε. Πάντως νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη η συνεισφορά μας στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ω σκιώδη λοιπόν εισηγητέ, θα είμαστε στη διάθεσή σα πολύ άμεσα για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα. Ευχαριστώ. Έχουμε και εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Έχουμε. Έχετε το λόγο. Δεν ήσασταν παρόν όταν μίλησε ο εισηγητή. ήρθατε να μας πείτε αυτά που σας έχουν γράψει. Δεν πειράζει, πείτε τα. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που καθυστέρησα λιγάκι, αλλά να πω ότι μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία, Ποιο είστε, Βίτο Μπορέλη από την Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, υπεύθυνο για τα προγράμματα Erasmus Mundus δεν ακούμε την πρόεδρο εκτός μικροφώνου. Well, ε, ε, ε, do you hear me? Με ακούτε? Δεν είμαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγώ. Είμαι από την σχετική υπηρεσία, αλλά ας δώσω πρώτα το λόγο στον συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσει τη φωνή του σε αυτή τη συζήτηση. Δυστυχώ πάλι δεν ακούμε την Πρόεδρο. Εντάξει λοιπόν. Ε, και πάλι με συγχωρείτε. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεύθυνο για το πρόγραμμα Εράσμου Mundus. Να επεκταθώ λίγο σε σχέση με όσα υπόθηκαν στι προηγούμενε παρεμβάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την προσπαθή ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία, ενδιαφέρεται ιδιαίτερω να αυξήσει την συμμετοχή των γειτονικών χωρών από την, τα ανατολικά και το Νότο στα προγράμματά μα. Ήδη κάποια κονδύλια του προπολογισμού θα διατεθούν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτο, το Σεπτέμβριο του 2011, συγκεκριμένα 20 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε περαιτέρω δράσει κινητικότητα για τον ερχόμενο ακαδημικό χρόνο. Αυτό θα γίνει μέσω του προ 2 του προγράμματο Erasmus Mundus, που συγκεκριμένα επικεντρώνεται στι γειτονικέ χώρε. Περισσότερη χρηματοδότηση προβλέπεται για την ερχόμενη διετία του προγράμματος, δηλαδή τη διετία μετά την τωρινή φάση. Επίσης, πρόσθετη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα νεολαία σε κίνηση, προκειμένου να βελτιώσουμε την οικοδόμηση δυνατοτήτων στις γειτονικέ χώρες, καθώς και την αδελφοποίηση και τον πολιτισμό γενικότερα. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε την πρότασή μας για την επόμενη γενιά προγραμμάτων και προβλέπουμε να υπάρχει συγκεκριμένη δράση για τις χώρες της γειτονιάς μας, προσπαθώντας να συνδυάσουμε πιο αποτελεσματικά τη διάσταση της οικοδόμησης δυνατοτήτων που εκπροσωπούν τα προγράμματα 10 και αυτά που αφορούν τον πολιτισμό με τα προγράμματα Εράσμου Μούντο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι με τη δική σα στήριξη θα έχουμε στοχευμένε δράσει για τι γειτονικέ χώρε. Ευχαριστώ. Και τώρα εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι στηρίζω πλήρω εκ μέρου τη υπηρεσία μα την προσέγγιση σα. Βρίσκουμε ότι οι παρατηρήσει είναι όλε έγκυρε, εύστοχε και μπορούν να αυξήσουν την ε, προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία της ανακοίνωση. Τό μόνο μπορούμε να κάνουμε λοιπόν να στηρίξουμε την προσεκύσή σα. Αλλά Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να στηρίξουμε την προσέγγιση σα Αλλά γεγονο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να παίρνει από εμά τα κονδύλια για να κάνει αυτό που θα επιθυμούσαμε και σε αυτό θα ήθελα λίγο να επεκταθώ. Του χρόνου ε, μπορούμε να αυξήσουμε μόνο το πρόγραμμα Erasmus Mundus και για το μεθεπόμενο έτος. Και λίγα πράγματα από το πρόγραμμα για τη διαβίου μάθηση. Αλλά στην έκθεση του κυρίου Μιγκάλσκι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το μέλλον και να έχουμε ένα κείμενο που να λέει νέα προγράμματα πρέπει να ανοίξουν για την πολιτική γειτονία στην εκπαίδευση και την παιδεία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα τα πάρουν από το δικό μας προπολογισμό. Και σήμερα ε, το άνοιγμα για τα Δυτικά Βαλκάνια δεν μπαίνουν από τα δικά μας κονδύλια αλλά από το ΙΠΑ που είναι το προενταξιακό μέσο και τα μελλοντικά κονδύλια δεν ξέρω πώς θα βαφτιστούν αλλά όχι από το δικό μας προϋπολογισμό στο πρόγραμμα της διαβίου μάθησης μεγαλύτερα προγράμματα κινητικότητας να διευρυνθούν και να επεκταθούν. Λοιπόν, και τα δύο πρέπει να κάνουμε. Και για του χρόνου, αυτό που κάνετε, να δώσουμε προσοχή, αλλά επιπλέον, για το επόμενο πρόγραμμα, την προγραμματική περίοδο, να προβλέψουμε να συνδεθούν οι χώρες αυτές με τα δικά μας προγράμματα εκπαίδευσης και μορφωτικών ανταλλαγών. Εντάξει, έχουμε και τις δύο ιδέες τότε μέσα. Με παρακολουθείτε. Μάλιστα, ο εισηγητή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω, συμφωνώ. Συμφωνώ αυτά τα προγράμματα να είναι απόλυτα ανοιχτά, Πρόεδρε και ελπίζω ότι αυτό θα βρει στη σωστή θέση στη διατύπωση την τελική στο κείμενο και από πλευρά ΕΛΚ ε, ένα σκιώδη εισηγητή ε, έχει διοριστεί. Το καλωσορίζουμε αυτό για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να προχωρήσουμε με τη δουλειά. Ο διασυνοριακός χαρακτήρας σε συγκεκριμένα προγράμματα που αναφέρονται σε αυτή τη γνωμοδότηση και αυτός πρέπει να αντανακλάται η κυρία Πακ, η κυρία Ναντέλοβα αναφέρθηκε σε αυτό και σε σχέση και με τόσο πρόσωπο της Επιτροπής ε, με το πρόγραμμα Έρασμος και το πρόγραμμα Τέμπους. Όλες αυτές οι ιδέες, ε, οι προτάσεις αυτές ε, πρέπει να μπορέσουν να προχωρήσουν. Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και τα κονδύλια ώστε να υποστηριχθούν. Και η Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης υποστηρίζει και αυτή, αυτή την κατεύθυνση. Προσβλέπω στη συνεργασία μας παρόλο το πιεστικό χρονοπλαίσιο. Ελπίζω ότι θα τελειώσουμε έγκαιρα τη δουλειά μα. Ε, Σα ευχαριστώ. Τι ε, τροπολογίε τις αναμένουμε επίση στις 8 Σεπτεμβρίου που εκπνέει η προθεσμία κατάθεσής τους όπως όλες ε, για τις, τις υπόλοιπες εκθέσεις. 8 Σεπτεμβρίου εκπνοή προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών. Ευχαριστώ. Περνάμε στο 16. Τις αποφάσεις των συντονιστών τις επικυρώσαμε σήμερα το πρωί ήδη. Όλα τα άλλα θέματα τα οποία είχαμε χθε στη συνάντηση των συντονιστών υπάρχουν κάποια προβλήματα για αυτά. Όχι. Περνάμε στο 17. Διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα. Ούτε και αυτά υπάρχουν. 18. Επόμενη συνεδρία, συνεδρίαση 4 και 5 Οκτωβρίου. Οι συντονιστές θα συνέλθουν στις 12 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο Συντονιστέ, 12 Σεπτεμβρίου Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη πρωία. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Εύχομαι καλοδιάθετη και με μεγάλη ε, όθηση να επανέλθετε μετά τις διακοπές για τις δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή. Στο καλό, γεια σα. Ευχαριστώ και του Διερμηνεί και για εσά καλέ διακοπέ. Καλέ διακοπέ για όλου. Ευχαριστώ.